Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Με τη 15 λεπτή καθυστέρηση ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας, αλλά Δευτέρα είναι, συμβαίνει. Σε ό,τι αφορά την ημερήσια διάταξη, πώς υπάρχουν παρατηρήσεις? Καταρχήν να αναφέρω ότι μεταδίδεται από το διαδίκτυο συνεδρίασή μας. Έχουμε διερμήνει από και προς 16 γλώσσες και να περάσουμε στην έγκριση των πρακτικών της 29ης και 30ης Αυγούστου του 2018. Ε, θα ακολουθήσουμε την γνωστή διαδικασία. Και περάμε στο σημείο 4, την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ροντρίγκο Ντελαπουέρτα Μοντόγια, τον διευθυντή του γραφείου της ΦΑΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βέλγιο, επευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας διατροφής. Όπως θα θυμάστε, η Παγκόσμια μέρα διατροφής εορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου. Ε, γιατί το, τέτοια μέρα ιδρύθηκε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1945. Επειδή όμως φέτος δεν έχουμε προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση εκείνες τις μέρες, σκεφτήκαμε να γιορτάσουμε σήμερα αυτή την Παγκόσμια Μέρα Διατροφής. Με μεγάλη λοιπόν χαρά θα ήθελα να καλωσορίσω και πάλι το Διευθυντή του Γραφείου της ΦΑΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βέλγιο, τον κύριο Ροντρίγκο Τελαπουέρτα Μοντόγια. Να το καλωσορίσω θερμότατα συνεδρίασή μας. Από ό,τι γνωρίζετε, ο κύριος Δελαπουέρτα συμμετείχε πρόσφατα στη συνεδρίασή μας στις 17 Μαΐου και εκεί μας ε, μίλησε για το πρόβλημα της ρήπανσης του εδάφους ε, και μας ενημέρωσε για τα απορίσματα του Παγκόσμιου Σεμιναρίου για το θέμα αυτό. Σήμερα θα μας παρουσιάσει την έκθεση του 2018 της ΦΑΟ για την επιστηστική ασφάλεια και τη και τη διατροφή στον κόσμο, καθώς και την έκθεση της ΦΑΟ για την κατάσταση της γεωργίας ε, σε σχέση με τη μετανάστευση και την αγροτική ανάπτυξη. Οπότε σκεφτήκαμε ότι είναι μια λαμπρή ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων με τον εκπρόσωπο τόσο ε, έγκυρης και σημαντικής οργάνωσης. Επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω να, να σας ενημερώσω μάλλον ότι μετά από πρόσκληση του Προέδρου, του Διευθυντή της ΦΑΟ, του κ. Γκρατσιάνο Ντασίλβα, θα στείλουμε ad hoc κοινή αντιπροσωπεία των Επιτροπών Γεωργίας και Ανάπτυξης στο Παγκόσμιο Κοινοβουλευτικό ε, φόρουμ ε, στην Παγκόσμια Κοινοβουλευτική Διάσκεψη Κορυφή για την καταπολέμηση τη πείνα και του υποσυτισμού που θα λάβει χώρα στη Μαδρίτη στα τέλη του μήνα. Προκειμένου να παγιωθούν οι πολιτικέ δεσμεύσει για την υλοποίηση του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη υπαριθμών 2. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω τον κύριο Τελαπουέρτα, του εκπροσώπου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του εκπροσώπου των άλλων θεσμικών οργάνων που παρακολουθούν αυτή τη σημαντική συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Να καλωσορίσω φυσικά και τους ευρωβουλευτές, τους συνεργάτες τους, τους αντιπροέδρους της Επιτροπής μας και να δώσω το λόγο στον καλεσμένο μας, τον κύριο Ντελαποέρτα Παρακαλώ, κύριε Διευθυντά. Α, συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Δες, που είναι ο συντονιστής της ομάδας του ΕΛΚ, ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε. Χρησιμοποιώ το δικαίωμα που έχω εξ ονόματος όλων των παρόντων συναδέλφων να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μας σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Οπότε σας εύχομαι ό,τι καλύτερο να έχετε υγεία και επιτυχίες στην Προεδρία σας εδώ στην Επιτροπή μας. Oddaję panu, panu ευχαριστώ. Ε, happy birthday. Χρόνια πολλά κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω δύο εμβληματικές εκθέσεις της ε, Οργάνωση Τροφίμων ε, και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η πρώτη αφορά την κατάσταση της επιστηστικής ασφάλειας και της διατροφής στον κόσμο με, τα, με το ακρονίμιο SOFI που δημοσιεύθηκε πριν από τρεις εβδομάδες και θα σας δώσω και κάποιες προκαταρκτικές σκέψεις για τη δεύτερη έκθεση με το ακρονίμιο ΣΟΦΑ που αφορά την κατάσταση του, της γεωργίας και των τροφίμων που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί επίσημα. Η δημοσίευση θα γίνει επισήμως στις 15 Οκτωβρίου και Τέλος, όπως είπε και ο Πρόεδρος, πολύ ευχαρίστω να σας παρουσιάσω τη φετινή Παγκόσμια ημέρα της διατροφής. Πριν όμως ξεκινήσω, θα ήθελα να σας αναφέρω κάποιες ε, καλές ειδήσει, χαρμόσυνες ειδήσει. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, στι 29 και 30 Οκτωβρίου θα οργανώσουμε στη Μαδρίτη την, το, την πρώτη Παγκόσμια Κοινοβουλευτική Διάσκεψη κορυφή για την καταπολέμηση τη πείνα και του υποσυτισμού στη Μαδρίτη, όπω είπα με στόχο να προωθεί η πολιτική βούληση για να υλοποιηθεί ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης αριθμό 2, δηλαδή ε, να εξαλειφθεί η πείνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και χαίρομαι ιδιαίτερος που ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Σταγιάννη, θα συμμετέχει στη, μαζί με μια επίσημη αντιπροσωπεία κοινοβουλευτικών που θα εκπροσωπούν ε, τις δύο επιτροπές ε, Γεωργίας και Ανάπτυξης και θα λάβουν μέρος ε, σε αυτή τη σημαντική διάσκεψη κορυφής. Σε ό,τι αφορά την πρώτη έκθεση που σας ανέφερα, την κατάσταση της επιστηστικής ασφάλειας και της διατροφής με τα αρχικά σόφη, όπως θα δείτε στο φυλάδιο που σας φέραμε, δημοσιεύθηκε για δεύτερη συνέχεια χρόνια από τη ΦΑΟ, μαζί με, άλλους, με τέσσερις άλλους σημαντικούς οργανισμούς ε, των ΗΕ, κάτι που συνιστά ήδη επίτευγμα αυτή η συνεργασία μεταξύ των οργανισμών του, του ε, Δυστυχώ όμω δεν είναι ευχάριστα τα νέα τη έκθεση. 821 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο υποσυτίζονταν το 2017. Αυτό σημαίνει αύξηση κατά 17 εκατομμύρια σε σχέση με το 2016. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ένας στους εννέα συνανθρώπους μας είναι χρονίως υποσυτισμένος στον κόσμο. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό γιατί έχει αντιστρέψει την θετική τάση μείωση τη πείνα που διαπιστώναμε τα 15 τελευταία χρόνια και μόνο τα τελευταία τρία χρόνια αντιστράφηκε αυτή η θετική τάση. Και είδαμε αύξηση και πάλι τη πείνα παγκοσμίω. Με άλλα λόγια, επιστρέφουμε στα στοιχεία που είχαμε για την πείνα πριν από μία οκταετία. Θα συμφωνείτε μαζί μου ότι κάτι τέτοιο απαιτεί άμεση δράση από όλου μα, αλλά και κάποιε μακροπρόθεσμε επενδύσει από όλου επίση. Και θα πρέπει να εντείνουμε τι προσπάθειέ μα για να υλοποιήσουμε τον στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη για μηδενική πείνα, για εξάλληψη τη πείνα μέχρι το 2030. Αλλά αν συνεχιστεί αυτή η αντιστροφή τη θετική τάση, ε, έχουμε ξεφύγει από το δρόμο μα. Το δεύτερο ρήμα τη έκθεση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μεταβλητότητα του κλίματος και τις ακραίες καιρικέ συνθήκες. Αυτό είναι ένα από του παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην άνοδο της πείνας και έχουμε εντοπίσει τρεις βασικές αιτίες για την αύξηση της πείνα. Ο ένας είναι η μεταβλητότητα, η αστάθεια του κλίματος με τις ακραίες καιρικέ συνθήκες, το δεύτερο είναι οι ένοπλε σειράξει. και ο τρίτος λόγος είναι η οικονομική κρίση, η ύφεση. Αυτοί οι τρεις λόγοι, αυτοί οι τρεις παράγοντες συνυπάρχουν και ελεπιδρούν μεταξύ τους κάτι που συνήθως συμβαίνει, η κατάσταση μόνο μπορεί να ενταθεί και να επιδεινωθεί λόγω αυτού του συνδυασμού των αιτιών σε πολλές χώρες του κόσμου. Επανέρχομαι τώρα σε μερικά από τα βασικά πορίσματα και στοιχεία της φετινής μας έκθεσης. Σας έχουμε φέρει ένα έντυπο και αντίγραφα της πλήρους έκθεσης, αλλά και στις διαφάνειες μου στο PowerPoint έχω ένα link ε, που μπορείτε να βρείτε την έκθεση. Όπως είπα, το 2017, 821 εκατομμύρια άνθρωποι μας υποσυτίζονταν. Μια θετική τάση, αν κοιτάξουμε την πρώτη στήλη, την γαλάζια, αν μπορούμε να το κρίνουμε θετικό, είναι ότι ο υποσυτισμός των παιδιών κάτω των 5 ετών, η των παιδιών που είναι καχεκτικά ή ε, λιπόσαρκα, αυτός ο αριθμό μειώνεται συνεχώ τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, εξακολουθεί να είναι υψηλός. 22% των παιδιών κάτω των 5 ετών εξακολουθούν να είναι καχεκτικά, λιπόσαρκα και να υποσυτίζονται. Περίπου 151 εκατομμύρια παιδιά δηλαδή. Επίσης πολύ ανησυχητικό είναι ότι 38 εκατομμύρια παιδιά είναι υπέρβαρα παγκοσμίω, ενώ η παχυσαρκία των ενηλίκων αυξάνεται παγκοσμίω. 13% των ενηλίκων στον κόσμο είναι παχύσαρκοι και τα μεγαλύτερα ποστά παχυσαρκία εντοπίζονται στη Βόρεια Αμερική, αλλά όλο παραδόξως αυξάνονται ταχύτατα στην Αφρική και την Ασία, κάτι που δεν θα το φανταζόμασταν, θα ήταν αδιανόητο στο παρελθόν. Ταυτόχρονα και όλους παραδόξως στις ίδιες χώρες διαπιστώνουμε και υποσυτισμό των παιδιών και καχεξία παιδική, αλλά ταυτόχρονα ανεμία στις γυναίκες, παιδική παχυσαρκία ή υπέρβαρους ενήλικες και αυτές οι πολλαπλές μορφές υποσυτισμού μπορεί να συνεπάρχουν όχι μόνο στην ίδια οικογένεια, αλλά και στον ίδιο άνθρωπο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ή στις διάφορες περιόδους της ζωής του. Όπως είπα και στην αρχή, ένας από τους ε, βασικούς παράγοντες και τα βασικά αίτια για την αύξηση της πείνας είναι οι ακραίες καιρικέ συνθήκες ε, ε, και οι κλιματικές αλλαγές. Όντως, το κλίμα έχει γίνει όλο και πιο ασταθές και μεταβλητό και οι ακραίες καιρικέ συνθήκες έχουν αυξηθεί και στη, στον αριθμό τους αλλά και στην έντασή τους. Και όπως βλέπετε στη γραφική παράσταση, η πάνω μοβ γραμμή που περιλαμβάνει τις περισσότερες κλιματικές αντικσότητες μας δείχνει ότι έχουμε κατά μέσο όρο 213 ε, ε, μέσες ή σημαντικές ε, φυσικές καταστροφές το χρόνο τέτοιου είδου ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικέ καταστροφέ ή θεομηνίε ε, συμβαίνουν κυρίω σε χώρε αγροτικέ, όπου ο πληθυσμό εξαρτάται από τη γεωργία. Και η αύξηση τη γεωργία, ε, το πλήγμα τη γεωργίας έχει αυξηθεί στι χώρε αυτέ. Θα πρέπει λοιπόν να καταστήσουμε τη γεωργία μας πιο ανθεκτική και ταυτόχρονα και βιώσιμη. Τα καλά νέα είναι ότι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε τη γνώση, έχουμε κάνει τη διάγνωση, έχουμε προγράμματα, έχουμε εργαλεία, έχουμε μηχανισμού στη διάθεσή μα για να βοηθήσουμε τον κόσμο και κυρίω του γεωργούς και κτηνοτρόφου να προσαρμοστούν και να προλάβουν τη μεταβλητότητα του κλίματο και τι ακραίε καιρικέ συνθήκε. Θέλουμε λοιπόν να παρατείνουμε κάποια προγράμματα, να τα διευρύνουμε, να διευρύνουμε τι πολιτικέ μα και να γίνουν πιο ανθεκτικέ στι κλιματικέ αλλαγέ. Και μάλιστα παγκοσμίω και καθ' όλη την αλυσίδα αξία τη γεωργία. Και μια και η επιστηστική ανασφάλεια είναι από του λόγου μετανάστευση, η μετανάστευση από την Ήπεθρο ε, είναι ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να σας επισημάνω. Και αυτό είναι το αντικείμενο της δεύτερης έκθεσης που σας ανέφερα. Στις 15 Οκτωβρίου, δηλαδή την παραμονή της Παγκόσμιας ημέρας διατροφής, θα δημοσιεύσουμε την έκθεση για την κατάσταση των τροφίμων και της γεωργίας. Η φετινή έκθεση θα διερευνήσει τις διασύνδεσεις που υπάρχουν μεταξύ ε, γεωργίας, αγροτικής ανάπτυξης και μετανάστευσης. Και μάλιστα θα δώσουμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τους ε, ηθήνοντες της πολιτικής. Σήμερα θα σας κάνω μια σύντομη επισκόπηση των βασικών ε, σημείων της έκθεσης και σας καλώ μετά τη δημοσίευση της έκθεσης να μας ε, στείλετε τις παρατηρήσεις αν επιθυμείτε. Καταρχήν διαπιστώσαμε ότι η εσωτερική μετανάστευση, η μετανάστευση στο εσωτερικό μιας χώρας είναι πολύ ευρύτερο φαινόμενο σε σχέση με τη διεθνή μετανάστευση. Δεύτερον, διαπιστώσαμε και έχουμε παρατηρήσει ότι η μετανάστευση μεταξύ των αναπτυσσομένων χωρών είναι πολύ ε, μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά το μέγεθός της από τη μετανάστευση μεταξύ από αναπτυσσόμενες προς ανεπτυγμένες χώρες στο πλαίσιο αυτό πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων κυρίως στις αγροτικές αλλά και στις αστικές περιοχές ε, των χωρών είναι βασική προτεραιότητα. Για παράδειγμα, η Αφρική θα πρέπει να παράγει 18 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης το χρόνο, να δημιουργεί 18 εκατομμύρια θέσεις εργασίας το χρόνο για να απορροφήσει τις νέες ε, εισόδους στην αγορά εργασίας. Ενώ μέχρι σήμερα η Αφρική μόνο 3 εκατομμύρια θέσεις, ε, επίσημες θέσεις εργασίας το χρόνο δημιουργεί. Δηλαδή 15 εκατομμύρια νέοι κάθε χρόνο ε, προστίθενται στο, συντελεστή, στο ποσοστό της ανεργίας στην Αφρική. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ένα μεγάλο τμήμα των διεθνών εμβασμάτων που στέλνουν εργαζόμενοι μετανάστες στις πατρίδες τους πηγαίνουν κυρίως προς τις αγροτικές περιοχές. Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι περισσότεροι μετανάστες ε, διεθνώς προέρχονται από αγροτικές περιοχές. Είτε πηγαίνουν στη γειτονική πόλη ή στη γειτονική περιοχή είτε στη γειτονική χώρα. Αλλά η μετανάστευση προέρχεται κυρίως από αγροτικές περιοχές. Αγαπητοί, συνα... αξιότιμοι ευρωβουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω να σας δείξω ένα βίντεο από την Παγκόσμια ημέρα διατροφής. As Όπως είδατε, το βασικό θέμα είναι οι δράσεις μας για, την, για το μέλλον και η εξάλληψη της ε, πείνας παγκοσμίω μέχρι το 2030 είναι εφικτή. Θέλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να υψώσουμε τη φωνή μας για να πούμε ότι είναι εφικτή η εξάλληψη της ε, ε, πείνας μέχρι το 2030, γιατί 80% των φτωχών παραμένουν στις αγροτικές περιοχές και ο βιοπορισμός ε, των συνανθρώπων μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γεωργία, την αλληλεία και τη δασοκομεία. Γι' αυτό η εξάλληψη της πείνας προϋποθέτει μετασχηματισμό της γεωργικής οικονομίας. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις στη γεωργία με σεβασμό των αρχών για τις υπεύθυνε επενδύσεις, να προωθήσουμε τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και να συνδέσουμε τους παραγού τροφίμων με τις αστικές αγορές. Η ΦΑΟ είναι έτοιμη να διαδραματίσει το ρόλο της και να συνεργαστεί με τους ηθήνοντες πολιτικής και με τις κυβερνήσεις, προσφέροντας ε, στατιστικά δεδομένα, στοιχεία, παρακολουθώντας τα δεδομένα αυτά και προσφέροντας συμβουλές για τη χάραξη ε, η προαγωγή και εφαρμογή διεθνών συνθηκών και νομικών πλαισίων προκειμένου να στηρίξουμε εθνικές στρατηγικές για τη γεωργία και τα τρόφιμα. Γι' αυτό καλούμε και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνεχίσουν, όπως έκαναν και στο παρελθόν, να μας υποστηρίζουν σε αυτή μας την προσπάθεια και σε αυτή το μας το ρόλο, γιατί και η δική σας συνεισφορά είναι θεμελιώδου σημασία. Και πραγματικά ε, ευελπιστώ αυτή η πρώτη παγκόσμια διάσκεψη κορυφής ε, ε, κοινοβουλευτικών ε, για την καταπολέμηση της πείνας και του υποσιτισμού, θα καταλήξει σε μια συνένεση των βουλευτών, των κοινοβουλευτικών παγκοσμίω για να υλοποιήσουμε έναν κόσμο χωρί πείνα και υποσυτισμό. Και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη αυτή τη Παγκόσμια Κοινοβουλευτική Διάσκεψη Κορυφή για την καταπολέμηση τη πείνα και του υποσυτισμού. Και να σα ενημερώσω για ένα άλλο, μια άλλη εκδήλωση που θα διοργανώσουμε στα πλαίσια τη ε, παγκόσμια ημέρας διατροφή. θα επικεντρωθούμε στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη για να υλοποιήσουμε το στόχο μα και να εξαλείψουμε την πείνα μέχρι το 2030. Αυτά σας ευχαριστώ και είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί σας. Η τελευταία διαφάνεια περιέχει τα στοιχεία μας που θα μας βρείτε, ε, το, την ιστοσελίδα μας, το λογαριασμό Twitter και είμαστε πρόθυμοι να συζητούμε όποτε επιθυμείτε τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση και φλέγον το ζήτημα για την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πραγματικά θεμελιώδης ο ρόλος της ΦΑΟ και πολύ σημαντική και η συνεργασία μας με την οργάνωση αυτή. Και θα συμμετέχουμε, όπως είπατε, στην διάσκεψη κορυφής της Μαδρίτης, που θα γίνει για πρώτη φορά σε τέτοιο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Περάμε τώρα στη συζήτηση. Το λόγο έχει πρώτο ο κύριος Νταντά. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτά που είπατε και που δείχνουν ότι το θέμα της πείνας στο κόσμο είναι θέμα προβληματισμού για πολλούς και θα πρέπει να συνεχίσει να είναι και για μας. Θα πρέπει να πάρουμε μέρος σε αυτή τη διαδικασία και να κάνουμε κάτι. Υπάρχει ένα θέμα στο οποίο δεν αναφερθήκατε. Το 2008-2009... Τα μέλη του G20 ζήτησαν από τη ΦΑΟ να αναλάβει μία αποστολή διαφάνειας των παγκόσμιων αποθερμάτων έτσι ώστε να μπορέσουν να καταπολεμήσουν την αύξηση των τιμών. Μπορείτε να μας πείτε πού ακριβώς βρίσκεται η ΦΑΟ. Οι τιμές ε, βεβαίως μειώθηκαν, ε, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν απασχολεί ιδιαίτερα την επικαιρότητα. Ο κύριος Δεκάστρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θερμά συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες για αυτή την ε, Ευχαριστούμε όλους τους εκπροσώπους της ΦΑΟ που συμμετείχαν σε αυτόν. Δυστυχώς είναι θέματα που μας αφορούν όλους και όπως έδειξαν οι γραφικές παραστάσεις που μας δείξατε, δίχως άλλο η κατάσταση βαίνει επιδεινούμενη και αυτό θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα της διατροφικής ασφάλειας και πόσο είναι υποχρέωσή μας να προωθήσουμε την ανάπτυξη σε συγκεκριμένες περιοχές της γης. Πρέπει να είναι πρωταρχικό μέλημα αυτό της Ευρώπης δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα μεταναστευτικά προβλήματα αν δεν αντιμετωπίσουμε θαραλέα και ευφυώς τα προβλήματα που πλήττουν τις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για ανάπτυξη. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε κοιτάζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζουν άλλες χώρες στον κόσμο. Ας δούμε πώς επενδύει η Κίνα. Στην Αφρική έγινε διάσκεψη σε μια, στη διάσκεψη κορυφής 50 αφρικανικών χωρών Γίνα παρουσίασε ένα πρόγραμμα επενδύσεων που ξεπερνούσε τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Το πρόγραμμα αυτό φορούσε την γεωρική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των υποδομών. Η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει κάτι περισσότερο και, αυτή η παγκόσμια διάσκεψη κορυφής στις 29 και 30 Οκτωβρίου θα μπορέσει να αυξήσει την ε, ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό της πείνας στον κόσμο. Εμείς ε, με τις ε, δυνάμεις μας εδώ στο Κοινοβούλιο θα γιορτάσουμε το World Food Aid. Υπάρχει και μια διαφάνεια. Στις 16 Οκτωβρίου θα γιορτάσουμε εδώ αυτή την, ε, με αυτή την ευκαιρία εδώ στο Κοινοβούλιο. 16 Οκτωβρίου και καλούνται βέβαια όλοι οι συνάδελφοι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά για την παρουσίασή σας. Κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία λέω στους γεωργούς ότι έχουν μια ευγενή αποστολή να τρέφουν τον κόσμο. Θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας σε ένα σημαντικό θέμα. Ο γεωργικός τομέας, όχι μόνο στη Ρουμανία αλλά και σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στην Ιρλανδία, βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα μεγάλο πρόβλημα, έλλειψη εργατικού δυναμικού. Είπατε ότι η ανεργία είναι πάρα πολύ υψηλή σε αυτό το κλάδο και Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ του να μπορέσετε να προσελκύσετε εργαζόμενους από άλλα μέρη του κόσμου και πραγματικά εμείς θα πρέπει να κάνουμε εισαγωγή εργατικού δυναμικού για να, μπορέσει να, μπορέσουν να επιβιώσουν οι αγρότες. Γιατί σήμερα μιλάμε για την καταγραφή των γεωργών, ενώ θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πάρα πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρόκειται να κλείσουν γιατί υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Κυρία Στράκερ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Μία συγκεκριμένη ερώτηση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ συχνά αναφερόμαστε το πρόβλημα του ασύλου, των μεταναστών, και αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία σε αυτά τα θέματα. Εμείς δεν πρέπει μόνο να μιλάμε, αλλά να βρίσκουμε και λύσεις, όπως είπατε πολύ σωστά. Θα πρέπει να δίνουμε μία ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους στην Ευρώπη. Αυτό που λείπει στην παρουσίασή σας είναι τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και να είναι κάτι απτό. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι πολύ συχνά οι γεωργοί και στη δική μου χώρα μου λένε έχουμε πολλές γνώσεις για να μπορέσουν να ξεκινήσουν διάφορα προγράμματα. Και οι γνώσεις αυτές κάπως θα πρέπει να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι στιγμή δεν έχουν γίνει και πάρα πολλά και πραγματικά δεν ξέρουν τι να κάνουν όλες αυτές τις γνώσεις. Κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Πρόεδρο του Γραφείου της ΦΑΟ για την παρουσίαση που μας έκανε. Όλοι γνωρίζουμε ότι το θέμα της εξάλληψης ε, της πείνας δεν είναι θέμα τροφίμων, αλλά θέμα πολιτικής. Και εμεί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε από του μεγαλύτερου δωρητέ στι αναπτυσσόμενε χώρε. Αλλά δυστυχώ τα χρήματα αυτά δεν καταλήγουν στα σωστά χέρια, ούτε εξυπηρετούν το σωστό σκοπό. Και μάλιστα από ό,τι ξέρουμε πρέπει να αυξήσουμε τον προπολογισμό κατά 17 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως για να φτάσουμε στα 100 εκατομμύρια ανθρώπων που απειλούνται από την πείνα. Πώς θα τα καταφέρουμε ε, και πώς μπορούμε σωστά να δρομολογήσουμε αυτά τα κονδύλια και που παρόλο που δορίζουμε δεν φτάνουν στα σωστά χέρια. Και σίγουρα δεν θα επιλύσουμε το πρόβλημα της πείνας αν δεν αντιμετωπίσουμε τις αιτίες της πείνας και ο στόχος της εξάλληψης της πείνας μέχρι το 2030 προϋποθέτει βιώσιμη γεωργία, βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη και ταυτόχρονα επίλυση των ενόπλων σειράξεων και ε, επίλυση όλων των αναπαραγόντων. 20 με 30 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται στα πρόθυρα, στο χείλος του θανάτου λόγω της πείνας, λιμοκτονούν τόσοι άνθρωποι. Και είπαμε ότι 800 εκατομμύρια άνθρωποι υποσυτίζονται ή 100 εκατομμύρια άνθρωποι κοίτονται στο κρεβάτι τους και δεν έχουν τι να φάνε. Αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ ενισχυτικές. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι απλά νούμερα, είναι ανθρώπινα πλάσματα, είναι ανθρώπινες ζωές και θα πρέπει να φροντίσουμε πολύ σοβαρά να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα μηνύματα και του εκτελεστικού διευθυντή του κυρίου Μπίσλι ότι θα πρέπει να συσπηρωθούμε, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά η πολιτική μας θα πρέπει να είναι σαφής και στοχευμένη και όχι όπως ήταν μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χόισλινγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά για την παρουσίασή σας. Πραγματικά μας παρουσιάσετε τα προβλήματα που δυστυχώς δεν λύνονται, αλλά αυξάνονται. Θέλω να σχολιάσω ένα θέμα, να, για να μου πείτε ποιες είναι οι πρακτικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Η Ευρώπη θεωρεί την Αφρική μια ε, μερική αγορά για τα προϊόντα τα αγροτικά. Πολλοί γεωργοί στην Αφρική δεν μπορούν να παράξουν ε, και η παραγωγή πραγματικά μειώνεται. Οπότε προφανώς πλήττονται πολύ περισσότερο οι ε, αγροτικές περιοχές. Κυρίως οι μικρές ε, εκμεταλλεύσεις, οι μικροί γεωργοί. Είπατε ότι υπάρχουν διάφορες περιφέρειες οι οποίες θα μπορούσαν να απτυχθούν. Πώς όμως ο ευρωπαϊκός δρόμος για να προωθήσουμε τέτοιου είδους περιφέρειες, ποιες είναι, τι είδους γεωργία θέλουμε να προχωρήσουμε, γεωργία με, υψηλά, με υψηλές τεχνολογικές προοπτικές, high-tech, με drones, ή θέλουμε τη γεωργία η οποία είναι βιώσιμη και η οποία είναι και οικολογική, βιολογική. Θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το μοντέλο που θέλουμε για την Αφρική, αντί να λέμε ότι πρέπει να, έχουμε μια γεωργία ε, υψηλής έντασης. Και επίσης αυτό που μας παρουσιάσατε και που είναι πάντα σαφές, δεν έχουμε λίγα τρόφιμα στον κόσμο. Θα μπορούσαμε να ταΐσουμε ουσιαστικά και 10 δισεκατομμύρια το κόσμο. Το θέμα είναι πώς κατανέμονται αυτά τα τρόφιμα και το θέμα είναι ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Και θα ήμουν ευγνώμων να μπορούσατε να μου απαντήσετε. Το θέμα δεν είναι να παράξουμε περισσότερα τρόφιμα, αλλά να, τα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται να κατανέμονται με σωστές και ε, δίκες προϋποθέσεις. «30% της ε, παραγωγής ε, στην Ευρώπη καταστρέφεται, αλλά το 30% αυτό δεν φτάνει ποτέ στην Αφρική γιατί λείπουν οι υποδομές». Νομίζω ότι κάτι και αυτό θα πρέπει να το συμπεριλάβετε στις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάιτς. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφο ο κύριο Χόσλινγκ και θέλω και εγώ να θέσω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Τι ακριβώ εννοείται με το μεγαλύτερε ιδιωτικέ επενδύσει στι αγροτικέ περιοχέ στην Ήπεθρο και επίση. Τι θα μπορούσατε, πώς θα μπορούσατε να συμβάλλετε στην, ε, στις διαπραγματεύσεις, ποια θα πρέπει να είναι η προλητική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Γεωργία, έτσι ώστε να καταφέρει όντως να μειώσει την πείνα στον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και για την παρουσίασή σας. Θα συνεχίσω στο ύφο ε, του συναδέλφου Χόισλινγκ, αλλά θα ε, επιλέξω μια διαφορετική κατεύθυνση στην Ευρώπη. Η διαφοροποίηση της γεωργίας είναι αυτή που, που, που αύξησε την ε, παροχή τροφίμων στην Ευρώπη, όταν δεν υπήρχε στην Ευρώπη επαρκής παραγωγή του. Το θέμα τώρα εδώ που θέτουμε είναι η εντατική γεωργία, η παραγωγή η βιώσιμη γεωργία, φιλική προς το περιβάλλον. Νομίζω όλα αυτά ε, μας εμποδίζουν να συμβάλλουμε στον αναπτυσσόμενο κόσμο, γιατί ουσιαστικά αγχωνόμαστε, ε, παρόλο που εμείς τρεφόμαστε πολύ σωστά, ενώ αυτοί που δεν τρέφονται χρειάζονται την τεχνολογία και λύσεις που να είναι βιώσιμες, που όντως να παράξουν τελικά αύξηση τροφίμων, να αντιμετωπίσουν τις ε, ζωονόσους, τις ασθένειες των φυτών και αυτό είναι μια πρόκληση ίσως και για μας μας. Ας αφήσουμε και εμείς τις, ε, κάποιες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε για τα συστήματα διατροφής μας εδώ στην Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο και ας δούμε λίγο περισσότερο τους ανθρώπους που έχουν όντως πρόβλημα στην Αφρική, ας τους δώσουμε φωνή. Γιατί πολλοί, ειδικά αν δούμε το θέμα της εργασίας και της τεχνολογίας, θέλουν να, να προχωρήσουν, θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη νέα τεχνολογία, αλλά η συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη νομίζω ότι πάει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι ε, για αυτούς τους τρεις ε, παράγοντες που αναφέρατε, που επηρεάζουν και δυσχεραίνουν την κατάσταση. Πρέπει να δούμε ποιος είναι ο μεγαλύτερος αντίκτυπος, γιατί σίγουρα οι συγκρούσεις είναι τεράστιο πρόβλημα και νομίζω ότι είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, ίσως κάποια ποσοστά, πόσο τους εκατό επηρεάζει το κλίμα, πόσο τους εκατό επηρεάζουν οι συγκρούσεις. Μιλήσατε και για την οικονομική επιβράδυνση, την κρίση. Και επίσης, ο υποσυτισμός δεν έχει να κάνει πάντα με την πείνα, πολύ συχνά έχει σχέση και με την παχυσαρκία, το είπατε κι εσείς. Οπότε πραγματικά προσβλέπω στις απαντήσεις σας και ε, περιμένω βεβαίως και την ε, ημέρα ε, διατροφής. Και όπως είπε και ο συναλφός υπάρχουν τρόφιμα. Το θέμα είναι ότι δεν κατανέμονται σωστά και αυτοί που δεν έχουν τα χρήματα να το αγοράσουν τελικώ είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν το σοβαρό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια. Γιατί είναι πραγματικά πολύ απογοητευτικό ότι πάνε 40 χρόνια από ό,τι θυμάμαι εγώ που ξεκινήσαμε να μιλούμε για το πρόβλημα της πείνας στον κόσμο. Και ενώ στις αναπτυγμένες χώρες καμαρώνουμε με την τεχνολογία μας και με τα επιτεύγματά μας, ταυτόχρονα δεν καταφέραμε να εξαλείψουμε μια δραματική, τραγική κατάσταση που οδηγεί ε, σε θάνατο εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο και προκαλεί τεράστια δεινά, οδύνη και νόσους, ασθένειες. Τι πήγε στραβά, πού βρίσκεται το πρόβλημα. Η ΦΑΟ αναλύει τα βαθύτερα αίτια αυτής της κατάστασης και ποια είναι αυτά τα βαθύτερα αίτια και οι βαθύτεροι λόγοι της πείνας. Και γιατί ήμασταν ανίκανοι να την εξαλείψουμε. Είδαμε ότι η επιστηστική βοήθεια κατέστρεψε χιλιάδες αγροκτήματα, μικρά αγροκτήματα στον κόσμο και οδήγησε σε αφανισμό τους μικροκαλλιεργητές. Επίσης είδαμε ότι ε, πριν έρθουν οι κανονισμοί για την ΚΑΠ, μας είπαν ότι ένας από τους στόχους μας ήταν να παράγουμε στην Ευρώπη τρόφιμα για να σητήσουμε τη, μέση τη μεσαία τάξη της Αφρικής, έτσι μας είπαν. Μήπως αυτός είναι ο λόγος που δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη της μικρής και μέσης γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, στις χώρες δηλαδή που πλήττονται από την πείνα και από τη συνέπειες της πείνας. Πιστεύω ότι αυτό είναι το βασικό αίτιο. Και αν δεν είμαστε ικανοί, αν ε, δείξουμε το θάρρος και την τόλμη να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, ελάχιστα θα σημειώσουμε πρόοδο. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω τι φάω και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η κατάσταση ότι αφορά την αγροτική μεταρρύθμιση, γιατί η φαρπαγή γεών και η επιβράδυνση της γεωρικής μεταρρύθμισης είναι ένα ουσιαστικό και, πραγμα... πολύ σοβαρό πρόβλημα. Επίσης, για τις κλιματικές αλλαγές. Είναι αναφυσβήτο ότι οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν τις εισοδίες και δημιουργούν προβλήματα αλλά δεν είναι αυτός ο μόνος λόγος, ούτε μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το πρόσχημα των κλιματικών αλλαγών για να ε, ε περιγράφω μια κατάσταση για την οποία φταίνει ο, κατα... καπιταλισμός και οι αναπτυγμένες χώρες εδώ και πολλά χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αγγιλέρα. Ευχαριστώ και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του Γραφείου της ΦΑΟ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία του και θα έχουμε την ευκαιρία και στη Μαδρίτη στα τέλη Οκτωβρίου να ανταλλάξουμε απόψεις, αλλά θα ήθελα να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Πιστεύετε ότι η Εμπορικέ συμφωνίες και οι συμφωνίες σύνδεσης που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αναπτυσσόμενες χώρες, για παράδειγμα τη βόρεια Αφρική επηρεάζουν προς το καλύτερο την κατάστασή τους, την πραγματική τους κατάσταση και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της έλλειψης τροφίμων που βιώνουν αυτές οι χώρες. Πιστεύετε ότι είναι προς όφελός αυτές οι συμφωνίες σύνδεσης και οι εμπορικές συμφωνίες ή απλώς ε, ή βελτιώνει την κατάσταση για τους Ευρωπαίους εισαγωγείς. Ερωτώ λοιπόν, ποιες είναι οι συνέπειες ε, των εμπορικών συμφωνιών και των συμφωνιών σύνδεσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις αναπτυσσόμενες χώρες και αν επηρεάζουν θετικά την επίλυση της πείνας και του υποσυτισμού. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους εκπροσώπους μάλλον, από τις Γενικές Διευθύνσεις Γεωργίας και Υγείας. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους εκπροσώπους ε, θέλει το λόγο. Πολύ ευχαριστώ. Τώρα. Α, δεν θέλετε. Καλώς. Οπότε μπορούμε να ξαναδώσουμε το λόγο στον Διευθυντή του Γραφείου της ΦΑΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βέλγιο για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Θα μπορούσατε επίσης να μιλήσετε και τις, την, την βιοτεχνική γεωργία, τη γεωργία μικρής κλίμακας. Γιατί και οι μικροκαλλιεργητές αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και οι μικροκαλλιεργητές ε, κυρίως ε, καλλιεργούν για την επιβίωσή τους. Επίσης, ανέκυψε το θέμα της ε, εντατικής γεωργίας κατά πόσο είναι χρήσιμη η αύξηση της παραγωγής. Επίσης, τι γίνεται με τις κινέζικες επενδύσεις στην Αφρική. Είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα και σε ποιο βαθμό εξυπηρετούν τα αφρικανικά συμφέροντα ή σε ποιο βαθμό εξυπηρετούν τα κινέζικα συμφέροντα, γιατί κάθε χώρα ασκεί πολιτική εξυπηρετώντας τα εθνικά της συμφέροντα. Τι γίνεται με τις κινέζικες επενδύσει λοιπόν στην Αφρική. Ευχαριστώ. Thank you very to... Ευχαριστώ όλους σας. Τώρα θα πρέπει να αρχιστώ στο πεδίο της μάχης. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σχεδόν σε όλα τα ερωτήματα. Ε, δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα, αλλά θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ο κύριος Ντατένα έκανε μία ερώτηση και η απάντησή μου είναι καταφατική. Το 2008, ναι, υπήρχε μία αύξηση της τιμής των τροφίμων στον κόσμο. Ακόμα θα έλεγα ότι ήταν στενά συνδεδεμένη αυτή η αύξηση με τις κλιματικές αλλαγές και έπληξε περισσότερο τους ε, ε, ανθρώπους με πενιχρά μέσα. Και βεβαίως ε, αυτοί που θίγονται περισσότερο είναι αυτοί που ζουν στις αγροτικές ε, περιοχές. Ήδη υπήρχε μια επιτροπή, αλλά έπαιζε ένα ελάσσονα ρόλο σε σχέση με το ρόλο που διαδραμάτισε μετά από 10 χρόνια. Στην ουσία υπήρχε συνεργασία με την κοινωνία των ε, πολιτών και το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει και μια ομάδα υπεύθυνων υψηλού επίπεδου που ελέγχουν το επίπεδο των τιμών. Θα πρέπει συνεπώς να δούμε αν παρατηρείται η αύξηση ενός συγκεκριμένου ε, είδους διατροφής. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε την Παγκόσμια Εβδομάδα της διατροφής θα γίνει μια συνάντηση που θα συμμετέχουν και πάρα πολλοί φορείς των Ηνωμένων Εθνών και όπως σας είπα, πολλοί εταίροι από διάφορους κλάδους. Σε ό,τι αφορά την παρέμβαση του κυρίου Ντικράτσιο σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι το Σάμιτ είναι μια μοναδική ευκαιρία, πρώτη φορά που οι βουλευτές από την Ασία, την Ευρώπη, η Λατινική Αμερική θα συναντηθούν προκειμένου να συζητήσουν πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Θα ήταν σκόπιμο αν θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τη συνάντηση αυτή για να καταλήξουμε σε μια γενική άποψη όλων των ευρωβουλευτών. Η βασική ιδέα θα πρέπει να είναι ότι όλοι θα πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας για την καταπολέμηση της πείνας στον κόσμο. Ο κύριος Ντεκάστρο είναι πρόεδρος της ε, Συμμαχίας δια ε, Κοινοβουλευτικής Συμμαχίας για την καταπολέμωση της πείνας. Ε, συμμετέχουν βουλευτές από όλες τις επιτροπές και πραγματικά ελπίζω και άλλα μέλη να μπορέσουν να πάρουν μέρος στη συμμαχία αυτή που είναι πάρα πολύ σημαντική για την καταπολέμηση της πείνας. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κυρίου Μπούντα, την έλλειψη δηλαδή εργατικού δυναμικού, ναι, έχετε δίκιο. Αν κοιτάξετε αντικειμενικά την Ευρώπη θα διαπιστώσετε ότι οι αγροτικές περιοχές χάνουν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους και χρειάζεται εργατικό δυναμικό. Υπάρχει η κυκλική προσωρινή μετανάστευση, η εποχική μετανάστευση. Έρχονται εργάτες για να βοηθήσουν και μετά επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Έχουμε αρκετά παραδείγματα υποστήριξης μεταναστών ή προσφύγων και στην Ευρώπη και σε όμορες χώρες. Ας πούμε συνεργαζόμαστε στενά με την τουρκική κυβέρνηση ε, και στηρίζουμε Σύριους ε, για να μπορούν να εργάζονται στο Γκαζιαντέπ. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη ε, για τις γυναίκες, αλλά εκεί έχουμε επιτύχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκπαιδευτεί και μπόρεσαν να απορροφηθούν από την αγορά της Τουρκίας. Και η τουρκική αγορά είναι ιδιαίτερα ε, ευτυχής. Εμείς λοιπόν διευκολύνουμε την ε, ένταξη των προσφύγων στις χώρες όπου βρίσκονται, γιατί δεν θα μείνουν εκεί για ένα μήνα. Θα χρειαστεί πάρα πολλής χρόνος για να τερματιστούν οι σειράξει στις χώρες τους. Έχουμε καλά παραδείγματα σε γειτονικέ περιοχές του Νοτιού Σουδάνα, που υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγες. Πάρα πολλοί πρόσφυγες πηγαίνουν για να εργαστούν σε αγροτικές περιοχές. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε ποια είναι τα αίτια, ποια είναι η ρίζα της μετανάστευσης, είναι αλλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τους πρόσφυγες που βρίσκονται σε άλλες χώρες, έτσι ώστε όταν επιτρέψουν στην γενέτειρά τους να έχουν, να έχουν αποκτήσει επιπλέον προσόντα και δεξιότητες. Έκανε μία ερώτηση ο κύριος Σρέτερ για τους ετούντες άσυλο. Νομίζω ότι απάντησα ήδη. Ε, παραθέτω στο παράδειγμα της ε, Τουρκίας ε, και των Σύριων προσφύγων. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να προωθούμε ιδέες και να διαδραματίζουμε κάποιο ρόλο για τους μετανάστες που βρίσκονται στην Ευρώπη. Έχουμε την οικονομία της γαλάζιας ελπίδας ε, για χώρες ε, της ε, Βόρειας Αφρικής. Για του κατοίκους που εργάζονται στον αλληλευτικό κλάδο. Όταν τα προβλήματα λυθούν στη χώρα τους μπορούν να επιστρέψουν. Έθεσε ένα ερώτημα και ο κύριος Πέτερ. Η κυρία Πέτε. Δεδομένα σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ε, τι ποσοστό οφείλεται στις κλιματικές αλλαγές, στις σειράξεις κτλ. Από τις 51 χώρες που βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρές κρίσεις, στις 37 υπάρχουν προβλήματα που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές. Είναι επίσης αλήθεια ότι οι χώρες όπως η Εμένη και η Σομαλία παρουσιάζουν και τα δύο φαινόμενα, και σειράξεις και κλιματικές αλλαγές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Όσο πιο πολλές μελέτες ε, κάνουμε, τόσο πιο εύκολα συνειδητοποιούμε πόσο ευάλωτος είναι ο κλάδος της γεωργίας, πόσο εξαρτώμενος από την ε, ε ίδρευση. Γιατί η ξηρασία είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα για τη γεωργία και από Γεωργία πλήττεται η Ανατολική Ασία, η Αφρική και ε, ο Γεωργός δεν μπορεί να παραμείνει και να καλλιεργήσει τη γη του. Όταν υπάρχει άρδευση, ε, υπάρχει ένα περιθώριο διάσωσης της γεωργίας. Σε περιπτώσεις, που, σε όμως που εξαρτώνται από τις ε, βροχοπτώσεις, Πολλοί γεωργοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη γη τους. Έγινε μια αναφορά στις αθέμητες πρακτικές, στις ενισχύσει και στην κοινή, κοινή γεωργική πολιτική. Στη ΦΑΟ πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επιτύχουμε ένα κράμα μεταξύ της βιοτεχνολογίας της αγροτεχνολογίας. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε κάτι που ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις. Πιστεύουμε ότι η βιοτεχνολογία είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει λοιπόν να συνδυάζουμε τις παραδοσιακές γνώσεις με την επιστημονική πρόοδο έτσι ώστε να μπορούμε να παράσχουμε επιστημονικές συμβουλές για σχετικά με το τι χρειάζεται κάθε χώρα. Έγινε μία αναφορά στην κοινή γεωργική πολιτική. Εμείς συμφωνούμε με τις συζητήσεις που έγιναν για τη γεωργική πολιτική, ιδιαίτερα ε, για θέματα συγχρονισμού της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής. Η αγροτική πολιτική είναι σημαντική προκειμένου να επιληθούν μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα. Οι τελευταίες προτάσεις της ΚΑΠ περιέχουν αναφορές ε, στην κατάσταση στον κόσμο, στη βιώσιμη γεωργία, στις κλιματικές αλλαγές, ε, στην περιβαλλοντική σταθερότητα, στην ε, άμβλυνση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η νέα αυτή πρόταση περιέχει αυτή την διεθνή πτυχή που μας βρίσκει σύμφωνους. Υπάρχει η σύνδεση μεταξύ των πάντων. Η γεωργία στην Ευρώπη συνδέεται με τη γεωργία ε, και σε άλλες χώρες. Έγινε μια αναφορά και στο εμπόριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη φάουνα ε, ασχοληθεί με το πώς θα μπορούσε να στηρίξει τις χώρες αυτές που βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο γιατί θα μπορούσε να προκύψει ένα όφελος και για τις νέες όμορες χώρες. Να μιλήσουμε και για την Task Force για την ε, Αφρική. Ε, είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Κομισιόν, διότι υπήρχαν κάποια, προ... ερωτήματα για το τι κάνει ο ιδιωτικό ε, τομέα και πώς μπορεί να βοηθήσει και πώς ε, τα αγροτρόφιμα και οι αγρο, αγροτικές ε, βιομηχανίες, εταιρείε μπορούν να βοηθήσουν και πώς μπορούμε να ε, ενισχύσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις στη Γεωργία στην Αφρική. Η Task αυτή ξεκίνησε να λειτουργεί το Μάιο, συναντάται τακτικά, συνεχίζει να κάνει τη δουλειά της. Νομίζω ότι αποτελεί ένα καλό βήμα για να αναλύσουμε το πώς ο ιδιωτικό τομέα μπορεί να συνεργαστεί για την Αφρική. Υπάρχουν κάποιε εθελοντακέ κατευθυντήρε γραμμέ ε, για τη διατήρηση γη, ε, για τι επενδύσει που είναι θεμελιώδου σημασία και ο ιδιωτικό τομέα ή η κινέζικη κυβέρνηση που αναφέρθηκε επίση πρέπει να τηρήσουν τους κανόνες αυτούς. Η Κίνα όλο και περισσότερο ε, προσπαθεί να τηρήσει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Ε, δεν είναι υποχρεωτικές φυσικά, είναι εθελοντικές, αλλά το θέμα είναι ότι έχουν ε, εγκριθεί από μια μεγάλη πλειοψηφία κρατών μελών και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει επίσης να τηρεί τους κανόνες αυτούς που απορρέουν από αυτές τις κατευθυντήριε γραμμές. Κυρίως όταν μιλούμε για τις ε, ευρωπαϊκές επενδύσεις, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το Εξωτερικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και αυτό, αυτός ένας τρόπος να επενδύουμε στον ε, γεωργικό τομέα, αλλά σεβόμενοι κανόνες. Μετά. Το ερώτημα για την ΚΑΠ ε, από τον κύριο Γουάλτς νομίζω ότι το, το απήντησα. Η τεχνολογία τώρα από την κυρία Μαγκίνες, ε, φυτο, ασθένειες των φυτών, ε, συνεργαζόμαστε όλο και περισσότερο με τον ιδιωτικό τομέα για να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους προβλήματα, να έχουμε καλύτερα δεδομένα, ώστε να παίρνονται καλύτερες αποφάσεις, να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για τους ε, γεωργούς. Το πρόβλημα το μεγάλο των ε, γεωργών στην Αφρική και των ε, αναπτυσσόμενων χωρών και στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ότι δεν θεωρούν ελκυστική τη γεωργία, ότι είναι κίνδυνος να επενδύσουν στη γεωργία. Δηλαδή η τεχνολογία και η σύνδεση υπαίθρου με, με αστικά κέντρα και αγροεταιρείες σημαίνει ότι θα πρέπει να παραμείνουν στις ε, ε, περιοχές αυτές εάν δούνε ότι ο γείτονάς τους πούμε, που έχει κάνει μια παρόμοια επένδυση θα πάει καλά. Ε, στις χώρες της Αφρικής όμως η γεωργία είναι πραγματικά θεμελιώδου σημασία τομέα, παρόλα αυτά εξακολουθεί να μην είναι ελκυστική για την νεολαία. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξουν ιδέε σκεπτικά για να μπορέσει ο τομέα τη γεωργία να γίνει και πάλι ελκυστικό. Παχυσαρκία σημαντικό θέμα για την Ευρώπη. 24% νομίζω των Ευρωπαίων είναι παχύσαρκοι, που είναι πραγματικά πολύ υψηλό ποσοστό και αυξάνεται. Η κατανομή τώρα των τροφίμων και παραγωγή τροφίμων πρέπει να παράξουμε περισσότερα τρόφιμα είναι σωστό ότι αν δει κανεί πόσα τρόφιμα πάνε χαμένα στον κόσμο, είναι το 1 τρίτο, 1,3 δις ευρώ δηλαδή. Μαθηματικά, με τους κανόνες, ε, με, με την ε, απώλεια τόσων τροφίμων θα μπορούσαμε όντω να έχουμε ταΐσει όλο τον κόσμο. Επίσης, είναι το πρόβλημα, της, το πρόβλημα δεν είναι μόνο της πρόσβασης. Στην υποσαχάρια Αφρική, ας πούμε, δεν υπάρχει παραγωγή τροφίμων, οπότε δεν μιλάμε για πρόσβαση εκεί. Και επίσης προσπαθούμε φυσικά να, ε, μειώνεται, να μειώνονται τα τρόφιμα που πετάγονται ουσιαστικά, να χρησιμοποιούμε καλύτερα τους φυσικούς πόρους, να σεβόμαστε τη βιοπικιλότητα, τα, τις γιές, Βεβαίω ο πληθυσμό αυξάνεται. Το 2050 θα έχουμε περίπου 10 δις πληθυσμό, αλλά και οι, ε, οι ροές και οι τρόποι κατανάλωσης επίσης ε, αλλάζουν. Ε, πολλοί καταναλώνουν φρούτα, κρέας που, που χρειάζεται για την παραγωγή τους πολύ περισσότερους φυσικούς πόρους. Οπότε πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ του να είμαστε μεν αυστηροί, το να εισάγουμε έστω και τα ελάχιστα, αλλά η ΦΑΟ υπολογίζει ότι πρέπει να παράξουμε 40 50% περισσότερα τρόφιμα μέχρι το 2050. Ε, προσπάθησα να απαντήσω στα περισσότερα ερωτήματα. Αν κάτι έχω ξεχάσει, ζητώ συγγνώμη. Σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες μας δώσατε και τις απαντήσεις στις απορίες των Ευρωβουλευτών. Και σίγουρα πολλές φορές μες τον Οκτώβριο θα εγγύψουμε σε αυτά τα θέματα. Γιατί έχουμε την έκθεση Δεκάστρο και την έκθεση πρωτοβουλίας. Και μην ξεχνούμε και στα τέλη, ότι στα τέλη ε, Οκτωβρίου θα έχουμε στη Μαδρίτη το Παγκόσμιο Κοινοβουλευτική Διάσκεψη Κορυφής, στην οποία θα συμμετέχουμε στην επίσημη αντιπροσωπεία που κινούμε την Επιτροπή ανάπτυξη. Και νομίζω ότι αυτή θα είναι ευκαιρία να επιστήσουμε την παγκόσμια προσοχή στα προβλήματα. Δηλαδή είναι παράδεκτο να έχουμε 800 εκατομμύρια και συνανθρώπου μα που υποσυντίζονται ή να έχουμε 30% σπατάλι τροφίμων, να πετάμε τρόφιμα. Ε, βέβαια η διατροφή αλλάζει, τα προβλήματα είναι πολλά, πολύ σύνθετα, αλλά σίγουρα το ζήτημα της διατροφής και της γεωργίας ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και είναι και το ζήτημα που κατεξοχή μας απασχολεί και στη συνεδριά της Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε λοιπόν κυρία Ντελαπουέρτα και σίγουρα θα έχουμε στενές επαφές και στο μέλλον, γιατί έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Και βρισκόμαστε και στο ίδιο μήκο κύματο ό,τι αφορά την επιτακτική ανάγκη να επιλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Σε ευχαριστούμε και πάλι. Και δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε κάνα δύο λεπτά ή αρκεί. Παρακαλώ. Τίποτα, μισό λεπτό. Θα ήθελα απλώ να σα ευχαριστήσω όλου θερμά για την πολύ καρποφόρα συζήτηση που είχαμε και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αμέριστη υποστήριξη που προσφέρει στη ΦΑΟ και για την προσπάθειά σας να καταστήσετε πιο βιώσιμη τη γεωργία και πιο φιλοπεριβαλλοντική. Σας ευχαριστώ επίσης για την προσοχή που δίνετε σε συγκεκριμένα θέματα όπως τα εδάφη, το νερό, το περιβάλλον και νομίζω ότι πολλά είναι τα επιτεύγματά μας την τελευταία δεκαετία. Δεν θα πρέπει να χάσουμε τη φόρα που έχουμε πάρει, την όθηση που έχουμε αποκτήσει και σίγουρα ε, είναι ανησυχητικά τα στοιχεία που έχουμε, αλλά θα μπορούσαμε να τα θεωρήσουμε ως ευκαιρία και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να εξαλείψουμε πραγματικά μέχρι το 2030 την πείνα παγκοσμίω. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ σημαντικό το μήνυμά σας, πολύ σημαντική αυτή η στόχη και μακάρι να καταφέρουμε να τους υλοποιήσουμε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τους εκπροσώπους. Παρακαλώ λάβετε θέση εδώ στο Προεδρείο για να μας παρουσιάσετε ε, την πρόταση για την αντιμετώπιση πολύ σοβαρού ζητήματος της ζωονόσου της Αφρικανικής Πανόλης των Χείρων. που δυστυχώς ε, απρόσμενα γρήγορα η επιζωτία αυτή έφτασε και στο Βέλγιο και πρόσφατα, πριν από καμιά δύο εβδομάδες, ο Βέλγος Υπουργός Γεωργίας ε, διέταξε τη σφαγή περίπου 4.020 των χείρων στην περιορισμένη ζώνη γύρω από την ε, περιφέρεια του, την επαρχία του Λουξεμβούργου που είχαν ασθενήσει με την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Αυτή η ζωονόσος πλήττει και τα οικόσιτα και τα αγριογουρούνα και εμφανίζεται στην Αφρική και τη Δυτική Ευρώπη. Μάλιστα κρούσματα αυτή τη στιγμή έχουν εμφανιστεί σε εννέα χώρες μέλη, Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία και Βέλγιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει κατά 50% στο κόστος κτηνιατρικής κάλυψης και βιοασφάλειας ε, σε σχέση με τα τρέχοντα μέτρα που εφαρμόζεται στο Βέλγιο και είναι έτοιμη να βοηθήσει όλα τα κράτη-μέλη προσφέροντας συμβουλές ή συγχρηματοδότηση για την καταπολέμηση της επιζωτίας. Πιστεύω όμως ότι καλύτερα θα μας τα πει ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΤΑ, της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ο κύριος Βαγκέτεμ, Μπέρναρ Βαγκέτεμ, πολύ συχνά έρχεται στην Επιτροπή μας. Μας έχει ε, απασχολήσει το θέμα γιατί έχουμε πολλά κρούσματα της επιζώτιας αυτής της χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Παρακαλώ, κύριε Βαγγέτα, με έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας κάνω μία επισκόπηση της κατάστασης. Ε, είχα έρθει και πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, στην Επιτροπή σας και έκτοτε είχαμε πολλές εξελίξεις, ενέσκυψαν πολλά περιστατικά και θα ήθελα να σας ενημερώσω για όλα αυτά. Καταρχήν θα σας παρουσιάσω την παρούσα κατάσταση της πρωτοβουλίας μετά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα τελευταία χρόνια, γιατί μην ξεχνάτε ότι πριν από τέσσερα χρόνια είχαμε ε, τα πρώτα κρούσματα αφρικανικής πανόλους των χείρων στις χώρες της Βαλτικής και τις πρώτες δράσεις. Θα ήθελα πρώτα να σας δείξω ένα σύντομο βιντεάκι που εξηγεί με σαφήνεια την κατάσταση. Βλέπετε τα πρώτα κρούσματα στη Γεωργία ή στη Ρωσική Ομοσπονδία και βλέπετε πώς έχει επεκταθεί η ζωονόσος το 2014 στη Ρωσική Ομοσπονδία. Σε όλη την επικράτη είχαμε κρούσματα και το 2015 είχαμε τα πρώτα κρούσματα στην Πολωνία και στις χώρες Βαλτικής. Βλέπετε τις πράσινες κουκίδες, θα σας εξηγήσω περί τι πρόκειται και βλέπετε την εξέλιξη μέχρι σήμερα που έχουμε πραγματικά μεγάλη κρίση ε, άριθμα κρούσματα. Είχαμε στη Ρουμανία, την ανατολική πλευρά της πολλά κρούσματα, κοντά στην, στον Εύξηνο Πόντο και μετά είδατε στη Ρωσία πώς επεκτάθηκε η ζωνόσος, αλλά και στην Ανατολική Ρωσία, πλησιάζοντας τα κινέζικα σύνορα που βρίσκονται εκτός του χάρτη της διαφάνειας, αλλά έχουμε ενημερωθεί ότι εδώ και ένα μισή μήνα είχαμε εκατοντάδες κρούσματα και στην Κίνα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε υποχρεωτική εξέταση και των αγριοχείρων. Οπότε όποιο αγριοχείρο βρίσκεται νεκρός εξετάζεται ε, για να ανοιχνευτεί η αφρικανική πανόλη των χείρων. Και οι περισσότεροι αγριόχειροι έχουν προσβληθεί. Γι' αυτό βλέπετε πολλές κουκίδες σε αυτό το τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι το ίδιο ισχύει και σε άλλε χώρε, τη Ρωσική Ομοσπονδία και την Ουκρανία. Αλλά εκεί δεν εξετάζονται οι αγριόχειροι για την ε, ζωνόσο αυτή. Εμείς ξέρουμε που βρίσκεται ο ιός, κάτι που δεν ισχύει για την Ουκρανία και τη Ρωσία. Γι' αυτό έχουμε διαπιστώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο ιός βρίσκεται και στους αγριόχειρους και βλέπετε τις πράσινες κοκκίδες για τους αγριόχειρους. Οι κίτρινες κοκκίδες είναι ε, χειροστάσια, εκτινοτροφικές ε, φάρμες και βλέπετε πώς εξελίσσεται η ζωονόσο στις χώρες της Βαλτικής. Ελάχιστες είναι οι φάρμες των χωρών της Βαλτικής που δεν έχουν μολυθεί. Έχουμε τις κίτρινες κουκίδες λοιπόν τα κρούσματα. Οι τελευταίες περιπτώσεις ήταν ε, στη, στο Βέλγιο μόνο για αγριόχειρους, αλλά έχουμε πάνω από 50 αγριόχειρους που έχουν ε, μολυνθεί και έχουν ε, εντοπιστεί και μάλιστα σε πολύ περιορισμένη ζώνη. Οι βελγικές αρχές λοιπόν με τα από Συμβουλή των Διεθνών Εμπειρογνωμόνων πρότειναν ε, μία ε, απαγόρευση κυκλοφορίας, ε, απαγόρευση εισόδου στο δάσος όπου βρέθηκαν οι μολυσμένοι αγριόχειροι. Η ίδια στρατηγική χρησιμοποιήθηκε και στην Τσεχία, όπου και εκεί είχαμε κρούσματα σε αγριόχειρους και εκεί χρησιμοποίησαν το ίδιο μέτρο, την ίδια στρατηγική και κατάφεραν να εξουδετερώσουν ε, την ε, ε, εξάπλωση της σου το τελευταίο εξάμεινο στην Τσεχία. Τώρα εκτός από τις χώρες τη έχουμε και την Πολωνία που έχει προσβληθεί από τη ζωνόσο. Έχουμε και το τρίγωνο Ουκρανία, Ουγγαρία και Ρουμανία. Και έχουμε και στο κέντρο της Ουγγαρίας μια, μια αιστεία, πάλι με αγριόχειρους και στην ανατολική πλευρά της Ρουμανίας είχαμε κρούσματα σε πάνω από χίλια χειροστάσια στη Ρουμανία και μία μονάδα κτηνοτροφική στη Βουλγαρία. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και θα επανέλθω στην κατάσταση στο Βέλγιο. Αυτός δεν είναι ο πρωινός χάρτης, αλλά χάρτης από την περασμένη εβδομάδα, δεν είναι σημερινός. Και βλέπετε το κόκκινο τμήμα είναι περιοχές που έχουν βρεθεί νεκροί αγριόχειροι στα δάση. Και το σημαντικότερο για να εμποδίσουμε την εξάπλωση της ζωνόσου είναι να ε, περισυλλέξουμε τους νεκρούς αγριόχειρους για να μην μολύνουν ε, άλλα ζώα. Γιατί για έξι μήνες παραμένει ενεργός ο ιός στο, στο σφάγιο, στο, ε, νεκρό αγριόχειρο. Γι' αυτό θα πρέπει να βελτιώσουμε τα μέτρα βιοασφάλειας και να μην αφήνουμε τους νεκρούς αγριόχειρους ε, ε, στο δάσος. Και βλέπετε σε, στην περιοχή που επιβλήθηκαν περιορισμοί και εκεί στο κέντρο βρέθηκαν οι μολυσμένοι νεκροί αγριόχειροι και απομακρύνθηκαν φυσικά από την περιοχή. Στη Βουλγαρία είχαμε ένα κρούσμα σε ένα χειροστάσιο και οι περισσότερες, τα περισσότερα μεμονωμένα κρούσματα οφείλονται στον ανθρώπινο παράδειγμα, όχι στην ε, αργή εξάπλωση της ε, ζωνόσου λόγω της μετακίνησης των αγριοχείρων. Εδώ οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα. Ε, έτσι μεταφέρθηκε ο ιός στη Βουλγαρία. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για πολύ δραστικό και επίμονο ιό και η Βουλγαρία εδώ και τις εβδομάδες ε, έχει καταφέρει να περιορίσει αυτή τη μόνη κτηνοτροφική μονάδα την ε, νόσο. Στη Ρουμανία βρίσκεται στην ανατολική πλευρά ε, τη συγκέντρωση και επίσης στη βορειοανατολική Ρουμανία έχουμε το δέλτα του Δούναβη, πολλά, πολλές, πολλά χειροστάσια και 20 τους χείρους σε αγροκτήματα και είναι δύσκολο και να συγκρατήσουμε την επέλαση και την εξάπλωση της νόσου. Βλέπετε πολλές πράσινες και κόκκινες κίτρινες κουκίδες και πολλούς αγριόχειρους. Οι ρουμανικές αρχές έχουν ε, σφαγιάσει πάνω από μισό εκατομμύριο χείρους το τελευταίο δίμηνο στη Ρουμανία για να αποφύγουν την εξάπλωση της ζωονόσου. Και από την άλλη πλευρά του χάρτη, στη γωνία με Ουγγαρία, Ουκρανία και Ρουμανία, έχουμε κάποια κρούσματα του ιού στα δάση, γιατί και έχουμε πυκνή ε, δασική περιοχή και είναι πολύ δύσκολο να περισυλλέξουμε τους νεκρούς αγριόχειρους. Α, τώρα, για το 2018, είχαμε, στη μία πλευρά έχουμε τα κρούσματα, τον αριθμό των κρούσματων και στην άλλη πλευρά τον αριθμό των ε, αγριοχείρων που έχουν περισυλλαγή. Τι έχουμε κάνει από την ε, αρχή του 2018 γιατί η κατάσταση ε, διαρκεί. Ήδη το 2014 έχουμε ασχοληθεί με το πρόβλημα που είχαμε τα πρώτα κρούσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Στέλνουμε λοιπόν εκεί την ε, ομάδα ε, κτηνιατρική εκτακτου ανάγκης ε, επιτόπου. Πρόκειται για εμπειρογνώμονες, ε, πραγματικούς εμπειρογνώμονες, κτηνιάτρου, όχι υπαλλήλου Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν υπάλληλοι απλοί. Στέλνουμε λοιπόν τους εμπειρογνώμονες και στείλαμε στι αρχέ του μήνα στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες και είναι εμπειρογνώμονε σε θέματα συμπεριφορά αγριοχείρων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί σε περιπτώσει όπω το Βέλγιο είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τι βελγικέ αρχέ να αντιληφθούν την κατάσταση. Και πρόκειται για κορυφαίου ε, διεθνεί εμπειρογνώμονε ε, που συμμετέχουν στο επιτελείο που στείλαμε στι βελγικέ αρχέ για παροχή συμβουλών μετά από τις εμπειρίες που είχαμε και στη Τσεχία αλλά και σε άλλες χώρες που έχουν πληγεί από τη ζωονόσο. Και βλέπετε δεξιά πώς κινούνται οι ε, κτηνίατροι στο δέλτα του Δούναβη, που είναι η διάζουσα η κατάσταση. Είναι 24 ώρες το 24ωρο διαθέσιμοι αυτοί οι εμπειρογνώμονες και έσπαψαν στο Βέλγιο λίγες ώρες αμέσως μετά την επίσημη ε, επιβεβαίωση των κρουσμάτων. Επίσης έχουμε επιθεωρητές που επανειλημμένως βρέθηκαν σε σύνορα ευρωπαϊκών χωρών με τρίτες χώρες και συμμετέχουν στην εγρήγορση μας ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των σύνορων για να αποφύγουμε παράνομες εισαγωγές κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξάπλωση τη νόσου όπω έγινε στο Βέλγιο και στη Τσεχία. Και είχαμε πολλέ αποστολέ σε θέματα, στα πλαίσια τη ετοιμότητας ε, που έχουμε, γιατί ξέρουμε θα φτάσει η ζωονόσος και θα εξαπλωθεί και χωρί την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Θα έχουμε επέκτασή της ένα με δύο χιλιόμετρα το μήνα. Οπότε είχαμε πολλές επιτόπιες απόστολες για να είμαστε σε ετοιμότητα και να ελέγξουμε την κατάσταση. Επίσης είχαμε μία πρωτοβουλία με τη μορφή της πλατφόρμας της ΦΑΟ, το GFTAT, Παγκόσμιο Πλαίσιο για την Εξάπληξη Διασυνοριακών Επιζωτιών. Είμαι μάλιστα πρόεδρος αυτής της ε, κοινή ομάδα της ΦΑΟ και του ΟΗΕ και επηρεάζει όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ε, συμμετέχουν όλες τις χώρες της Ευρώπης, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεδριάζουμε δύο με τρεις φορές το χρόνο για ανταλλαγή πληροφοριών και των πρακτικών. Την τελευταία συνεδρίαση την είχαμε στη Βαρσοβία. Εκεί εξετάσαμε πόσο σημαντική είναι η διαχείριση των αγριοχείρων και του περιβάλλοντος. Και βλέπετε... Ε, εδώ είναι μια φωτογραφία από την συνεδρίαση στη Βαρσοβία. Έχουμε, συζητήσαμε τη διαχείριση του κυνηγιού, γιατί είναι η υποστήριξη και η συνεργασία με τους κυνηγούς είναι θεμελιώδη σημασία για την καταπολέμηση της ζωνόσου. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι τη σημασία που έχουν οι βέλτιστες πρακτικές και να τις εφαρμόσουν στις ε, περιοχές που έχουν πληγεί από παλιά έχουν πληγεί τελευταία ή ακόμη δεν έχουν εμφανίσει κρούσματα. Αλλιώ δεν πρόκειται χωρί τη συνεργασία των κυνηγών να εξαλείψουμε την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Σε ό,τι αφορά τι ε, περιοχέ που εξακολουθούν να ε, μην έχουν εμφανίσει ε, κρούσματα, επαναλαμβάνω και χωρίς τη συμμετοχή του ανθρώπου η επέκταση της νόσου θα γίνεται κάθε μήνα ε, με ταχύτητα 1 με 2 χιλιόμετρα το μήνα. Λόγω της μετακίνησης των αγριοχείρων θα πρέπει να μειώσουμε την πυκνότητα αγριοχείρων, του πληθυσμού αγριοχείρων σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Μόνο έτσι θα μειώσουμε την, ε, την πιθανότητα να εξαπλωθεί περαιτέρω η επιζώτια. Αυτό λοιπόν που ήταν πάρα πολύ σημαντικό ήταν τι να κάνουμε με τα ε, σφάγια και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ασφάλεια κατά τη διάρκεια του κυνηγιού. Στις ε, βαλτικές ε, χώρες οι κυνηγοί δεν ε, χρησιμοποιούν σωστές πρακτικές βιοασφάλειας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να αποφευθεί μια περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Συζητήσαμε με υπουργού από τις χώρες όπου υπάρχει παρουσία της νόσου, διοργανώθηκαν αρκετές συνεδριάσεις. Έγινε μια σημαντική συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις αρχές Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια στρατηγική τώρα με βάση την εμπειρία μας, με βάση την εμπειρία των εμπειρογνωμόνων. Διαμορφώθηκε λοιπόν αυτή η στρατηγική η οποία αναθεωρείται από τους εμπειρογνώμονες. Τη βλέπετε εδώ. Αφορά την απαγόρευση στάθμευσης τους, ε, ε, με συγχωρείτε, τη δημιουργία ε, διαχωριστικών στους ε, αυτοκινητοδρόμους και άλλα μέτρα. Τι ακριβώς κάνουμε στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά την περιφερειοποίηση. τι κάνουμε με τις χώρες μέλη. Δώσαμε έναν περιφερειακό χαρακτήρα, υπάρχουν τρεις περιοχές οι κόκκινες περιοχές είναι οι περιοχές που έχουν υπάρξει ε, κρούσματα σε αγροκτήματα. Οι ροζ περιοχές ε, εμφανίστηκαν περιστατικά μόνο στα ελεύθερα ζώα και οι μπλε περιοχές είναι διάμεσες περιοχές όπου επιβάλλουμε περιορισμούς. Στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν κάνουμε τίποτα και κάναμε αυτή την περιφερειοποίηση για να μπορέσει η εσωτερική αγορά να συνεχίσει να ε, δραστηριοποιείται. Έχουμε λοιπόν τις χώρες της Βαλτικής, η βορειοτοκή πλευρά της Πολωνίας, ένα μέρος της Ρουμανίας, Τσεχία και εκεί υπάρχουν περιορισμοί, σύντομα θα έρθουν. Και έχουμε και μία μικρή κίτρινη περιοχή στη Βουλγαρία και μία άλλη στο νότιο ε, Βέλγιο. Και βεβαίως υπάρχει πάντοτε η Σαρδινία όπου υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια η νόσος. Το σημαντικό στοιχείο εδώ είναι η περιφερειοποίηση η οποία επικαιροποιείται κάθε φορά. Θέλουμε οι περιοχές της Ευρώπης που είναι απαλλαγμένες της νόσου να παραμείνουν ως έχουν και να μην επιμολύονται από άλλες. Έχει γίνει πολλή δουλειά και από την ΕΦΣΑ. Εδώ βλέπετε την γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ. Η Επιτροπή άρχισε να απευθύνεται στην ΕΦΣΑ πολύ καιρό πριν εμφανιστεί το πρώτο κρούσμα της νόσου. Τώρα είμαστε εν αναμονή της νέας γνωμοδότησης της ΕΨΑ, γνωμοδότηση η οποία ήταν ε, πάρα πολύ χρήσιμη στο τέλος της χρονιάς και πάλι η γνωμοδότηση αυτή για την επιδεολογική αξιολόγηση θα υποβληθεί σε μερικές εβδομάδες ή μήνες και έχουμε και μία γνωμοδότηση σε ΕΦΣΑ σε ό,τι αφορά την πυκνότητα των αγριόχειρων. Δηλαδή, μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να φτάσουμε για να μην υπάρξει εξάπλωση της νόσου. Η ΕΦΣΑ δυστυχώς δεν μπόρεσε να ορίσει ένα κατόφλι, δηλαδή ε, πόσο θα πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός των αγριόχειρων. Ε, η ΕΦΣΑ είναι της άποψης ότι τα διαχωριστικά, οι φράχτες δεν είναι πάρα πολύ χρήσιμοι για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Τώρα, οικονομική υποστήριξη, όπως είπε και ο πρόεδρος ε, στην ε, αρχή, εμείς υποστηρίξαμε οικονομικά τις ζώνες που είχαν πληγεί από την νόσο. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ετοιμότητας, συνεργαστήκαμε με την Ουκρανία και με την Μολδαβία και χρηματοδοτούμε και καμπάνιες ευαισθητοποίησης όχι μόνο στις χώρες μέλη που έχουν πληγεί αλλά και στις χώρες που είναι ελεύθερες της νόσου. Τώρα υπάρχει μια ε, πρωτοβουλία, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι η περιφερειοποίηση είναι επαρκής ε, και, να έχουμε τη βεβαιότητα ότι συνεχίζει να υφίσταται η εσωτερική αγορά. Έχουμε απαγορεύσει την ε, ε, μεταφορά αγριόχειρων σε άλλες χώρες. Δεν ε, δόθηκαν εξαιρέσεις για την ε, εγγραφή χείρων εδώ και δύο χρόνια. Χρηματοδοτούμε για την ανάπτυξη εμβολίων, ο μόνος τρόπος εκρίζωσης της νόσου θα είναι μέσα από την χρήση ενός εμβολίου, ό, μιλάμε για στοματικό χορηγούμενο εμβόλιο. Θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρό πριν αναπτυχθεί αυτό το εμβόλιο και να αρχίσει να χρησιμοποιείται στο δάσος. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρξει μία εξτρατεία ευαισθητοποίησης. Η εξαρτήσει αυτέ χρηματοδοτούνται και στις ε, χώρε που δεν έχουν πληγεί από την όσο. Εμείς προσπαθήσαμε να οργανώσουμε πολλές δράσει, αποκινούμε τους κυνηγού και τους γεωργούς, γιατί χωρίς την υποστήριξη των κυνηγών δεν θα μπορέσουμε να εκριζώσουμε την όσο και θα πρέπει να υπάρξει και μία αύξηση της βιοασφάλειας προκειμένου να μην ε, πληγούν τα αγροκτήματα ο ανθρώπινος παράγοντας, καθοριστικός ο ρόλος του στην διάδοση της νόσου στην Βουλγαρία, στην Τεχία, μερικές φορές και στην Πολωνία. Εκεί καταβάλουμε μια προσπάθεια να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για να αποφευθεί η διάδοση της νόσου και βεβαίως το θέμα της βιοασφάλειας. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά σε όλα τα αγροκτήματα. Θα πρέπει να δούμε τώρα ποια είναι τα επόμενα βήματα, αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια. Αυτά θα συναντηθούν ε, στο ε, στη συνάντηση Αγκριφής 15 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία με περιβαλλοντικά ε, ιδρύματα. Θα πρέπει να σταλεί μια επιστολή, έχουμε τη συνδιάσκεψη 19 Δεκεμβρίου και εμείς θα συνεχίσουμε να εμπλέκουμε τους κυνηγού και για το λόγο αυτό προβλέψαμε μία διοργάνωση με την ΦΕΙΣ που είναι η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση ε, Κυνηγών. Ε, μπορείτε βεβαίως να βρείτε περαιτέρω στοιχεία στην ιστοσελίδα που σας παρέθεσα. Ελπίζω να μην μακρηγόρησε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να ακούσουμε τώρα τους βουλευτές που θέλουν το λόγο. Τόμ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Κύριε Φαχούτεμ, η κατάσταση με, τον, ε, με την Αφρικανική Πανόλη των Χείραων στο Βέλγιο είναι ιδιαίτερο οξία. Αλλά βεβαίω αυτό ε, επεκτείνεται και σε άλλε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρία ερωτήματα θέλω να θέσω, που ίσω να είναι σημαντικά Καταρχάς, το θέμα του ανθρώπινου παράγοντα. Πάντα λέμε ότι η ε, διάδοση μιας ε, νόσου ε, μπορεί να οφείλεται και στον ανθρώπινο παράγοντα. Υπάρχουν ε, διάφορες εφήμες, ας πούμε ένας ε, ε, οδηγός φορτηγού πέταξε ένα υλικό που ήταν μολυσμένο ή πήγαν να κυνηγήσουν οι κυνηγοί σε μέρος που είχε κρούσματα. Ξέρετε για ποιο λόγο ξαφνικά βρέθηκε στο Βέλγιο η ζώνος αυτή. Ποια είναι η αιτία. Μετά, τα μέτρα βιοασφάλειας που αναφέρατε. Έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις βελγικές αρχές συνεργάζεται πολύ καλά. Εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε η συνεργασία να συνεχίζεται απρόσκοπτα. απρόσκοπτα. Αλλά οι γεωργοί ε, φυσικά ε, λαμβάνουν πολύ σοβαρά τα όσα γίνονται και το θέμα είναι τι γίνεται με τους αποστολείς. Ας πούμε, τα φορτηγά που πάνε από τη μία χώρα στην άλλη. Μήπως πρέπει και αυτοί να μπουν στην όλη διαδικασία. Και ένα ερώτημα για την Τσεχία. Υπήρξαν κάποιες ειδήσει που έλεγαν ότι οι τσεχικές αρχές ε, επιβάλλουν ε, επιπλέον ε, ελέγχους στο χείριο κράση από το Βέλγιο. Ε, μένα με εξέπληξε αυτό, γιατί για τα ε, γιατί για κάποια είδη χείρων ε, δεν έχει διαπιστωθεί ε, η ζωονόσος. Οπότε αυτό η έξτρα δηλαδή η έλεγχοι δεν θα επηρεάζουν την ιστορική αγορά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή της. Νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ καλά τα όσα γίνονται. Αυτό που ακούω που ε, επιτόπου ε, φωνές ε, λένε ότι ε, η Κομισιόν έχει όντως ε, δράσει άμεσα. Θα συμφωνήσω με τον Βέλγο συνάδελφο και θέλω και εγώ να ρωτήσω ποια ήταν η αιτία για αυτή τη γρήγορη επέκταση της ζωονόσου. Δεν είναι φυσιολογική αυτή η ταχύτητα. Καλό θα ήταν λοιπόν να έχουμε μια εξήγηση. Και μετά, πώ μπορούμε να φροντίσουμε ότι όταν υπάρχουν τέτοια κρούσματα θα μπορέσουμε να έχουμε περιορισμό των, ε, του απεριορισμού του αντικτύπου. Θεωρείτε ότι τα κράτη-μέλη είναι οπλισμένα όπως πρέπει για να μπορέσουν να λάβουν έξτρα μέτρα πούμε για να αποφύγουμε περαιτέρω διεύρυνση, επέκταση της, ασθεν... της ε, για να μην ε, περάσει από τους αγριόχειρους ας πούμε ε, στους ε, χείρους για ανθρώπινη κατανάλωση. Ο κύριος Ντός. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Αφρικανική Πανόλη των χείρων είναι πραγματικά μεγάλη πρόκληση για όλη την Ευρώπη. Ε, βρίσκονται κρούσματα αυτή τη στιγμή σε 10 ε, κράτη-μέλη. Εμείς στην Ουγγαρία καταφέραμε να αποφύγουμε ε, να επηρεαστούν ή να ασθενήσουν οι δικοί μας χείροι. Λάβαμε τα απαραίτητα μέτρα. Η Τσεχία, στην Τσεχία και στο Βέλγιο μόνο στους αγριόχειρους διαπιστώθηκαν τα κρούσματα της νόσου. Ε, προφανώς πρέπει να υπάρξει προστασία και επίσης πρέπει να αποζημιώσουμε τους ε, ε, γεωργούς, τους κτηνοτρόφους. Πρέπει να υπάρξουν τα απαραίτητα κονδύλια δηλαδή. Διάφοροι συνάδελφοι και εγώ ε, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε 15 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς γι' αυτό, για τους κτηνοτρόφους. Η Κομισιόν λοιπόν στις διαπραγματεύσει θα πρέπει να στηρίξει και την, ε, αυτή την πτυχή για, την, ε, για τον προπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Επίσης, η Κομισιόν θα πρέπει να δει και τις τρίτες χώρες, την Κίνα, την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ θα πρέπει να πείσει αυτές τις χώρες ότι η αρχή αυτή της περιφερειοποίησης θα πρέπει να γίνει αποδεκτή και από αυτές. Και δεν θα πρέπει να έχουν μια συνολική απαγόρευση λόγω της αφρικανικής πανόλης των χείρων. Θα πρέπει, αν θέλουν να απαγορεύσουν, να απαγορεύσουν μόνο τις, ε, τα, τα μέρη στα οποία όντως υπάρχει κρούσμα της ασθένειας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ε, παρουσίασή σας. Βλέπουμε και στο χάρτη που μας δείξατε ότι η Ρουμανία είναι αρκετά κόκκινη. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέτυχε να διαχειριστεί αυτό το πρόβλημα. Το 2014 εγώ σας έλεγα ότι υπάρχει κίνδυνος στην ε, Ρουμανία ακριβώς επειδή υπήρχαν δύο ε, κρούσματα ήδη στα ανατολικά της χώρας δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς, ε, μου είπε ότι ε, όλα είναι υποέλεγχο, ότι θα μας βοηθήσετε. Όντως μας βοηθήσατε, αλλά δεν, δεν παρενέβητε, βοηθήσατε τα κράτη-μέλη, αλλά δεν ε, κάνατε συγκεκριμένους ελέγχους, ας πούμε, να δείτε τι γίνεται στα κρατη αυτά. Και γι' αυτό η χώρα είναι σχεδόν ολοκόκκινη δεν ελέγξατε τον αριθμό των ε, χείρων, έγιναν πολλές συζητήσεις για το πόσα, ε, πόσοι χείροι ένα εκτάριο θα πρέπει να εκτρέφονται. Γιατί δεν παρενέβητε για να εξασφαλίσετε ότι όντως ο πληθυσμός των χείρων θα ελέγχεται. Οι αγριόχειροι τώρα, ε, τα άγρια ζώα, είναι σημαντικό. Η Ρουμανία έχει περίπου 60% του πληθυσμού των αγριόχειρων στην Ευρώπη. Έχει περισσότερους λύκους επίσης από την υπόλοιπη Ευρώπη και δεν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε γιατί απαγορεύεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Τι θα κάνουμε λοιπόν με το πρόβλημα αυτό, με αυτή την ασθένεια. Η αυτή η ασθένεια είναι χειρότερη και από τον έμπολα σε σχέση με τα όσα μας λένε οι, κτηνίατροι. Αλλά αν δεν έχουμε ολοκληρωμένα συνολικά μέτρα για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την ασθένεια αυτή, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα τελικά. Και οι συνάδελφοι ρωτάνε πώς έφτασε στο Βέλγιο αυτή η ερώτηση. Πολύ καλή, αυτή η ασθένεια. Πολύ καλή ερώτηση. Και υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα στη Ρουμανία. Τα ηχείρια αυτή Θάβονται στο χώμα, στη γη. Δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι κίνδυνος είναι αυτός. Ο ιός μένει δηλαδή στο χώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά μπορεί να έρθει ας πούμε μέσω κάποιου τροκτικού στην επιφάνεια, από κάποιο ε, υπόγειο ή από μια λεπού. Τι κάνετε λοιπόν για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη ας πούμε να ε, αγοράσουν ε, ε, συστήματα καύσης αντί να, να, να καίνε τα μολυσμένα, τους μολυσμένους χείρους αντί να τους θάβουν. αν λοιπόν δεν τα έχουμε όλα αυτά υπόψη μας και δεν λάβουμε έγκαιρα μέτρα θα καταλήξουμε και στο μέλλον σε παρόμοια κατάσταση. Και κλείνω. Πολλοί από τους κτηνοτρόφους αναρωτιούνται τι γίνεται στο ανατολικά της Ευρώπης. Έχουμε προβλήματα στην Ουγγαρία, έχουμε προβλήματα στη Βουλγαρία, έχουμε προβλήματα στη Ρουμανία και πολλοί από τους δυτικούς γεωργούς αναρωτιούνται τι κάνουν στην Ανατολική Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να περάσετε από το να, να βοηθάτε τα κράτη-μέλη στο να παρεμβαίνετε περιοχέ φορές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο συνάδελφος. Και εσείς ως ε, Κομισιόν ε, μιλήσατε για προβλήματα και οικονομικά, αλλά βεβαίως πρέπει να δείτε και το πρόβλημα των ακτινοτρόφων που έχουν πληγεί από την ε, ε αυτή. Είχαμε και στις κάτω χώρες την δεκαετία του 90 ε, τέτοια ζωνόσο και από τότε συζητούμε πώς θα το αποτρέψουμε στο μέλλον. Μιλήσαμε και για τους λύκους. Υπάρχει ένας λύκος που σκοτώνει έναν αγριόχειρο και μπορεί να κινηθεί ε, όχι μόνο 5 χιλιόμετρα, 155 χιλιόμετρα. Άρα θα εξακολουθήσει και αυτός να αποτελεί κίνδυνο. Και επίσης, τι γίνεται με, τις, ε, με τους πληθυσμούς αγριοχείρων. Ε, μπορούν κάτι να κάνουν τα κρατημέλη και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν την ε, ζωονόσο. Και επίσης, οι εμβολιασμοί. Έχουμε τα μέσα για να γίνουν εμβολιασμοί. Γίνεται υπερκής έρευνα προς αυτό. Γιατί δεν μιλούμε περισσότερο για εμβολιασμούς ούδη, ήδη θα έπρεπε να έχουν ληφθεί τέτοιου είδου αποφάσει. Και επίση ε, κάνετε παρεμβάσει κι εσεί, αλλά εγώ έχω ένα ερώτημα. Ε, σύντομα, πολλοί ε, ε, κυνηγοί θα ξεκινήσουν να κυνηγούν. Έχουμε κάτι για να ελέγξουμε τι θα γίνει στις περιοχές που θα κυνηγήσουν, οι οποίες έχουν ίσως πληγεί από τέτοια κρούσματα, γιατί μιλούμε για εκατοντάδες κυνηγούς που θα πάνε σε όλη την Ευρώπη. Πώς μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη Γενική Διεύθυνση Υγείας για την παρουσίαση. Πριν από ένα χρόνο είχα θέσει ένα ερώτημα για συγκεκριμένα μέτρα. Είχα ζητήσει να ληφθούν μέτρα. Εν τω μεταξύ τα πράγματα πήγαν καλά με την ε, ε, με τα στοιχεία που έχουμε είδαμε ότι η, οι ε, ε, ε, κυνηγοί πρέπει όντως να, να μπουν στην όλη διαδικασία εκπόνηση αυτού του εγχειριδίου. Αυτό που δεν έγινε καλό, δεν έγινε σωστά όμως, είναι οι περιοχές ξεκούρασης στους αυτοκινητοδρόμους. Και κάτι άλλο που λείπει είναι τι γίνεται με την εκπαίδευση με των συμφεροντούχων ή των υπαλλήλων οι ανησυχίες των γεωργών είναι πολύ σημαντικές ακόμα και σε χώρες που δεν έχουν πληγεί από την ζωνόσο. Οπότε και εκεί θα πρέπει να προχωρήσει η εκπαίδευση. Ως προς αυτό τι κάνουμε. Δύο ερωτήματα επίσης. Για τα ε, ε, κράτη-μέλη που επλήγησαν και που έχουν ε, αριθμό κρουσμάτων υψηλό έχουν υπάρξει οποιασδήποτε δηλώσεις ότι ας πούμε είναι, ε, μειώνονται τα κρούσματα. Τα μέτρα, όπως ας πούμε είχαμε εμείς στην Βαβαρία πέρσι, είχαμε, πάνω από, ε, είχαμε σκοτώσει πάνω από 90.000 αγριόχειρους ακριβώς για να, προλάβουμε τον κίνδυνο. Και για μένα είναι επίσης σημαντικό η συνεργασία με τα κράτη όπως η Ρωσία, πώς λειτουργεί υπάρχει κάποια κοινή γραμμή, υπάρχουν ε, συνεργασίες, ε, συνεργατισμοί, οτιδήποτε, γιατί νομίζω ότι μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει αυτή την ε, ζωονόσο και επίσης δεν έχουμε και εμβολιασμούς, οπότε τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Μόνο μέσω συνεργασίας με την Ρωσία ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ευχαριστώ. Η κυρία presidente. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σημαντική η παρουσίαση που μας έκανε ο εκπρόσωπος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να σας ε, διαβεώσω ότι με ανησυχεί πολύ η κατάσταση. Μας είπατε ότι με το θέμα αυτό έχω, ασχολούμαστε από το 2010 με στοιχεία και ανάλυση. Και παρόλα αυτά είδαμε εξάπλωση της σου και αύξηση των κρουσμάτων ε, και επέκταση σε πολύ περισσότερες χώρες. Είχαμε ακόμη και στο Βέλγιο τελευταία κρούσματα. Πώς είναι δυνατόν να ασχολείστε με το θέμα αυτό τόσα χρόνια και παρόλα αυτά να μην έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε την εξάπλωση της ε, ζώνος. Πού οφείλεται αυτό. Οι χώρες φταίνε που δεν έχουν εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα. Γιατί αυτή η αποτυχία στον έλεγχο της επιζωτίας. Γιατί αντί να έχουμε περιορισμό έχουμε αύξηση και εξάπλωση σε όλο και περισσότερες χώρες. Η δική μου πατρίδα, η Ισπανία, έχει πολλά, πολλούς χείρους. Οπότε η κατάσταση μας επηρεάζει. Τι μέτρα πιστεύετε θα πρέπει να ληφθούν που δεν έχουν ληφθεί ακόμη, ακόμη και από τις χώρες που δεν έχουν εντοπίσει ακόμη κρούσματα της επιζώτιας αυτής της Αφρικανικής Πανόλου των Χείρων. Ευχαριστώ κύριος Νταντά. Ευχαριστώ. Πριν από δύο χρόνια, δεν κάνω λάθος, είχατε έρθει για να μας παρουσιάσετε τους κινδύνους ε, της άγριας πανίδας για την δημόσια υγεία και την γεωργική οικονομία. Και δύο χρόνια μετά, δυστυχώς, έχουμε και την ε, γρήπη των πουλερικών, ε, μας είχατε έρθει στο παρελθόν και σήμερα την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων που επηρεάζει το χειροτρόφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω δύο ερωτήσεις. Αναφερθήκατε στο θέμα του εμβολίου που δεν είναι ακόμη έτοιμο. Υπάρχουν ελπίδες όμως. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που μας δίνουν κάποιες ελπίδες ή το θέμα του εμβολιασμού είναι ακόμη ένα ουτοπικό όνειρο. Και δεύτερο, μας είπατε για το σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουν οι κυνηγοί στην διαχείριση του πληθυσμού των αγριοχείρων που ε, εμφανίζεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης και η πυκνότητα, πυκνότητα του πληθυσμού αγριοχείρων είναι μεγάλη. Ε, θα πρέπει ίσως εμείς να ασκούσουμε κάποιες πιέσεις ε, στις οργανώσεις κυνηγών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ασχοληθεί με αυτό. Κύριε Σκούσμιουκ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διεξοδική ανάλυση που μας έκανε του προβλήματος. Κάθε μήνα η κατάσταση επιδεινώνεται δυστυχώς και έχουμε ήδη καμιά δεκαριά χώρες που έχουν πληγεί. Και μάλιστα το Βέλγιο, παρόλο που βρίσκεται μακριά από τις προηγούμενες αισθήσεις, έχει πληγεί και αυτό από τη ζωονόσο. Και ευχαριστώ και για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις ε, διάφορες χώρες. Βέβαια τα 60 εκατομμύρια που έχετε προβλέψει για υποστήριξη σε τέσσερα χρόνια είναι κάποια υποστήριξη, αλλά είναι μικρό το κονδύλιο. Δεν ε, ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα του φαινομένου. Και νομίζω ότι χώρες όπως η Πολωνία δικαιούνται λόγω της ε, έκτασης της ζώνης πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη. Υπάρχει δυνατότητα αύξηση. Επίσης, στην Πολωνία τα τελευταία τέσσερα χρόνια είχαμε αισθητή ε, πρόοδο σε ό,τι αφορά την εξάπλωση της νόσου και μάλιστα τελευταία είχαμε κάποιες ε, ριζοσπαστικές αποφάσεις ό,τι αφορά τους ε, αγριόχειρους και ακόμη και η κυνηγή που μέχρι τώρα ήταν σε ό,τι αφορά την εξάλληψη του πληθυσμού των αγριοχείρων, τώρα θα λαμβάνουν ε, βραβεία σημαντικά ε, χρήματα για να σκοτώνουν αγριόχειρους και ελπίζω ε, χάρη στη συμμετοχή και στα βραβεία τα οικονομικά έπαθελα που θα δίνουμε στους κυνηγού ε, να καταφέρουμε να περιορίσουμε στα, το πληθυσμό των αγριοχείρων. Αναφερθήκατε και στο θέμα των εμβολίων, του εμβολιασμού. Έχω την αίσθηση ότι είναι όνειρο απατηλό, ε, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον, το θέμα των εμβολιασμών. Δεν ξέρω σε τι φάση της έρευνας για την ανάπτυξη του εμβολίου βρισκόμαστε. Είστε σε θέση να μας πείτε πότε ακριβώς θα περιμένουμε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο για την όσο αυτή. Ευχαριστώ κυρία Σένερα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, τι ελέγχους κάνετε στα, στους αγριόχειρους, στις χώρες που είναι προς το παρόν ε, απαλλαγμένες από αφρικανική πανόλη των χείρων. Τι μέτρα έχετε λάβει για να αποφύγετε την εξάπλωση του ε, πληθυσμού αγριοχείρων και αυτών των χωρών. Επίσης, ε, ε, ψάχνετε και για άλλε νόσους στου αγριόχειρου, τη φυματίωση για παράδειγμα, για να αποφύγουμε πιθανή επιμόλυση και των βοηδών από τους αγριόχειρου σε άλλες νόσους όπως, ή σε νόσους όπως η σε η φυματιωση Ευχαριστώ. Βλέπω ότι δεν έχουμε δανεική διερμήνη, οπότε θα αναγκαστώ να μιλήσω αγγλικά. Θα ήθελα καταρχά να μου πείτε ποια, σε ποια συμφωνία έχετε καταλήξει. γιατί ακούω ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση για τους φράκτες. Ε, στη Δανία έχουμε 30 εκατομμύρια χείρους και θέλουμε να μπει ένας φράχτης μεταξύ της Δανίας και της ε, Γερμανίας που να καλύπτουν 75 χιλιόμετρα. Η Επιτροπή μας κατέστησε σαφές ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα φράχτη, πρέπει να προφυλάξουμε τους αγρότες μας. Επίσης, πέστε μου τι κάνετε σε ό,τι αφορά τα φορτηγά ε, αν προέρχονται από χώρες στις οποίες παρουσιάστηκαν κρούσματα, τι γίνεται. Ενδεχομένως ε, μεταφέρουν ε, την νόσο. Τι κάνει η Επιτροπή γι' αυτό. Και τι συμφωνία έχετε κάνει με τους κυνηγούς. Μπορούν να κυνηγήσουν σε μία περιοχή και να μετακινηθούν σε μία άλλη χωρίς να καθαρίσουν τα ρούχα τους ή τις ε, μπότες τους. Νομίζω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει και να καταλήξει σε ορισμένες συμφωνίες. Γι' αυτό το ερώτημά μου είναι τι είδους συμφωνίες έχετε συνάψει, τι έχετε σκοπό να κάνετε. Θα ήθελα και πάλι να σας ρωτήσω πότε κατά την άποψή σας θα ολοκληρωθεί το εμβόλιο. Το θέμα είναι να έχουμε δεδομένα, να μην περιοριζόμαστε σε μία απλή αναφορά. Έχω μία παράκληση, αγαπητοί συνάδελφοι. Αν έχετε ερωτήσεις, ε, να τις κάνετε τώρα και όχι απλώς να αναφέρετε παρατηρήσεις, γιατί έχει πτήσει, πρέπει να φύγει για την Αυστρία σε λίγο ο καλεσμένος μας. Οπότε παρακαλώ, μισό λεπτό και μόνο ερωτήσεις. Γιατί πριν, πριν από λίγο μόνο μου είπε ότι πρέπει να φύγει γιατί πετάει για Αυστρία και έτσι δεν μπόρεσα να ρυθμίσω από την αρχή το χρόνο. Ο κύριος Χόισλινγκ, παρακαλώ. Μισό λεπτό. Θα προσπαθήσω. Ε, τα ερωτήματα τα έθεσαν οι συνάδελφοι. Ε, υπάρχουν πολλοί ε, λόγοι να αρνηθεί κανείς ε, να κάνει κάτι, αλλά τώρα να χρησιμοποιούμε τα, τους χείρους για να το κάνουμε, πρέπει να δείτε στην ακρόαση τι μας είπατε. Είπατε ότι αν, γίνεται, αν υπάρχει έτσι εντατικό κυνήγι θα υπάρξει και μεγαλύτερη ε, επέκταση της, ε, της νόσου. Και τι θα γίνει δηλαδή, θα περιμένουν οι κυνηγοί να πεθάνει ο ιός για να βγουν να κυνηγήσουν. Δεν είναι λίγο δεν είναι ξεκάθαρο αυτό που μας λέτε. αν μπορείτε να μας το διευκρινίσετε. Ε, ότι αφορά την ε, προστασία των αυλών. Σε ό,τι αφορά τις, ε, τους οικόσιτους χείρους, τι ακριβώς κάνει η Ευρώπη. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ερώτημα αυτό, γιατί εγώ προέρχομαι από μια περιοχή που ήταν από τις πρώτες που επλήγησαν από αυτό το πρόβλημα. Χρειάστηκε να θάψουμε πάνω από 24.000 χείρους και πραγματικά δεν καταφέραμε να καταλάβουμε από πού προήρθε το πρόβλημα. Από μία, δύο, τρία αγροκτήματα και δεν έχουμε καταλάβει τα αίτια. Και επειδή δεν γνωρίζουμε τα αίτημα, το ερώτημά μου είναι πώς μπορούμε να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε αυτό το θέμα. Το δεύτερο ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να περιορίσουμε την έλευση μολυσμένων αγριόχειρων από την Λευκορωσία. Ε, ε, εμείς βρίσκουμε μια λύση στο πρόβλημα και ε, συνεχίζουν να έρχονται ζώα. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου καταρχάς να αναφερθώ σε μερικά συγκεκριμένα ερωτήματα που ετέθησαν από αρκετά μέλη. Σε ό,τι αφορά τους πόρους, τους οικονομικούς πόρους, στην δική μας ε, περιοχή έχουμε το κτηνοτροφικό πρόγραμμα και το, το πρόγραμμα, το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης ε, γίνονται, δίνονται αποζημιώσεις για τα ζώα τα οποία θανατώνονται. Θα Αυτή είναι η οικονομική πόρη που δίνουμε κατ' ουσία στις ε, χώρες μέλη. Εμείς αποζημιώνουμε για το 50%. Στα πλαίσια του κτηνιατικού προγράμματος προσαρμόσαμε τα μέτρα που είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση κατά 50%. Μερικές φορές μπορεί αυτή η χρηματοδότηση να φτάσει στο 75%. Και εγώ ανέφερα προηγουμένως ότι ένα από τα βασικά θέματα είναι η ανάκτηση των νεκρών μολυσμένων χείρων από το, χείρων από το δάσος. Πολλές ε, ε, χώρες μέλη έχουν εφαρμόσει προγράμματα που προβλέπουν την ε, αμοιβή ανθρώπων που αναζητάν νεκρούς ε, αγριόχειρους στα δάση και αυτό προκειμένου να αποφευθεί μια περαιτέρω εξάπλωση της νόσου και εμείς προσπαθήσαμε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε ε, εξτρατείες ευαισθητοποίησης υπάρχει και μια καμπάνια που θα πρέπει να γίνει από τις χώρες μέλη προκειμένου να υπάρχει βεβαιότητα ότι τα άτομα που ε, ταξιδεύουν από την Ανατολική Ευρώπη, όχι μόνο από την Ένωση, έχουν απόλυτη συνείδηση του, των κινδύνων που συνεπάγεται η εξάπλωση. Η δική μας συμβολή μεταξύ των άλλων είναι με ερευνητικά προγράμματα ύψους 40 ε, εκατομμυρίων ευρώ, ε, ε, προγράμματα ερευνών στον, για, την ανέβρεση, για το εμβόλιο. Είναι σαφές ότι στο εγγύς μέλλον δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί η έρευνα για το εμβόλιο. Οι έρευνες αυτές γίνονται εδώ και πολλά χρόνια. Ξέρετε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, είναι εμπολισμένη η Σαρδινία. Είναι πολύ δύσκολο όμως να βρεθεί το εμβόλιο. Κανένα δεν μπόρεσε να, βρεθεί, να βρει ένα αποτελεσματικό ε, εμβόλιο. Αν σε 10-20 χρόνια υπάρξει ένα εμβόλιο, το πρώτο θα είναι νέσιμο βεβαίως, και δεν ξέρω αν θα ε, ε, μπορεί κανείς να το δώσει στους ε, αγριόχειρους. Εμείς καταφέραμε να εκριζώσουμε την λύσα γιατί ακριβώς βρέθηκε εμβόλιο. Φαντάζομαι ότι τα επόμενα 30 χρόνια δεν θα υπάρχει εμβόλιο για τους αγριόχειρους. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε να ζούμε ε, με την ε, νόσο. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει η εκρίζωση της νόσου. Η ΕΦΣΑ ε, δεν μπορούσε να μας ορίσει ένα κατόφλι. Δεν μπορεί κανείς να ανατώσει όλους τους αγριόχειρους, δεν είναι ρεαλιστικό αυτό, δεν μπορεί απλά και μόνο να γίνει. Δεν μπορούμε να εγκριζώσουμε ούτε όλους τους αγριόχειρους, ούτε όλα τα πουλιά. Εμείς ε, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε για τα επόμενα 20-30 χρόνια με την Αφρικανική Πανόλη ε, των ε, χείρων. μια μεγάλη περιοχή του πλανήτη έχει προσβληθεί από την Πανόλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους φράκτες, ένα θέμα που έθιξαν αρκετοί από εσά. δεν θα βοηθήσουν οι φράκτες ε, που καλύπτουν μια μεγάλη απόσταση. Και αυτό σε ό,τι αφορά την μετάδοση της νόσου. Οι ε, αγλιόχειροι μπορούν να περάσουν από πάνω από τους φράκτες, από κάτω από τους φράκτες, να βγουν στον αυτοκινητόδρομο. Ε, όχι, είναι λανθασμένη η αντίληψη ότι μπορεί κανείς να αποφύγει τη διάδοση της νόσου με φράκτες. Στην Τσεχία μπήκαν μικροί ε, φράκτες. Ενδεχομένως θα τοποθετηθούν και στο Βέλγιο. Αυτό είναι κάτι εφικτό. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ετοιμότητας, όλα τα κράτη-μέλη είχαν άμεση εμπλοκή στα όσα κάναμε αυτά τα χρόνια για να αυξηθεί η ετοιμότητα. Δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός, τις βοηθήσαμε, ε, οργανώνονται εργαστήρια, διεθνείς ε, συναντήσεις και οι χώρες που έχουν ε, προσληθεί μοιράζονται τις γνώσεις τους με χώρες που δεν έχουν ακόμα προσληθεί. Πώς θα διαδοθεί η νόσος, σας είπα ότι αν εφαρμόσετε όλα τα μέτρα που συνιστώνται από τους ειδικού, η νόσος θα διαδοθεί ένα-δύο χιλιόμετρα το μήνα. Αν κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, σημαίνει ότι υπησέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Δηλαδή η διάδοση δεν οφείλεται στη φυσική ε, μετακίνηση των αγριόχειρων αλλά σε μηχανισμούς που επιτρέπουν στον ιό ε, να διαδίδεται με μεγαλύτερη ευκολία. Θα ήθελα να παραθέσω το τέταρτο παράδειγμα που είχαμε στην Βουλγαρία, την ε, Ουγγαρία, την Τσεχία. Εκεί έγινε ένα άλμα της νόσου. Εκεί αυτό οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα, όχι στη μετακίνηση του αγριόχειρου. Κατά κάποιον τρόπο ο ιός έφτασε εκεί διαμέσου ενός ανθρώπινου παράγοντα. Κάποιος άνθρωπος ε, το μετέφερε με τα παπούτσια του, με μολυσμένο κρέας. Υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρόποι ε, για να εξηγηθεί η επιδημιολογία της νόσου ο Βέλγος συνάδελφος έκανε μία ερώτηση σχετικά με το πώς εισήχθη η νόσος στο Βέλγιο. Όχι, δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε στοιχεία, δεν ξέρουμε πώς πέρασε η νόσος αυτή ε, στο Βέλγιο. Πολύ φορβάμε ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ε, εντοπίσουμε το πώς και το πότε πέρασε η νόσος στο Βέλγιο. Το θέμα είναι η συνεργασία με τους ε, κυνηγού. Αν δεν ανακαλύψουμε νωρί την ε, νόσο θα έχουμε περαιτέρω ε, κρούσματα και περαιτέρω διάδοση. Όταν ανακαλύπτει κανείς την νόσο θα πρέπει να γίνει προσπάθεια αποφυγής, απαγόρευσης του κυνηγίου. Μόλις λοιπόν ε, προσβληθεί ένα ζώο πεθαίνει μέσα σε 5-10 μέρες. Αν αφήσουμε το δάσος ως έχει χωρίς να ενοχλούμε τους ε, αγριόχειρους, οι αγριόχειροι θα πεθάνουν και εσείς από την πλευρά σας θα πρέπει να έχετε τη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει διάδοση της νόσου αλλά θα πρέπει επίσης να κάνετε κάτι και με το νεκρό ε, ζώο προκειμένου να μην διαδοθεί και άλλο η νόσος. Υπάρχουν περισσότεροι αγριόχειροι τώρα από ό,τι ήταν υπήρχαν στο παρελθόν και θα πρέπει, θα έλεγα, να γνωρίζουμε επακριβώς πόσοι αγριόχειροι υπάρχουν στην περιοχή. Αυτό όμω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ θα ήθελα να σας παραθέσω ένα παράδειγμα στο περίφημο δάσος στην Ιεχεία. Υπολογίστηκε ότι υπάρχουν 200 250, ε, αγριόχειροι. Αυτό το, τον εμβολιασμό τον έκαναν οι καλύτεροι εμπειρογνώμονε. Μετά όμω βρέθηκαν 650 νεκροί αγιόχειροι. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι να γίνουν εκτιμήσεις. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι φέτος έχουμε περισσότερους αγριόχειρους από ποτέ. Τι κάνουμε για να, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη. Προσπαθούμε να τους ε, παρέχουμε την απαραίτητη ε, ε, πρόσβαση στους εμπειρογνώμονες και να τους δίνουμε στοιχεία για να μπορούν να ελέγχουν την όσο Τώρα, και πάλι θα ήθελα να σας δείξω το χάρτη της Ευρώπης. Εμείς εφαρμόσαμε την περιφερειοποίηση, την ε, διαχωρισμό αναπεριφέρειες, επιτυχώς, επιτυχώς, έτσι ώστε η περιοχή ελεύθερη της νόσου να παραμείνει ελεύθερη της νόσου. Υπάρχουν ορισμένες ε, τρίτες χώρες, ε, τις οποίες συμπεριλαμβάνουμε σε αυτή την ε, αυτό το χωρισμό αναπεριφέρειες, άλλες χώρες δεν συμπεριλαμβάνονται όπως η ε, Ρωσία για παράδειγμα. Και το πάνελ που συναντήθηκε επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ καλά έκανε που εφάρμοσε αυτή την αρχή της ε, διαχωρισμού αναπεριφέρειες και ελπίζουμε να μπορέσουν οι τρίτες χώρες να εκμεταλλευτούν αυτή τη διαδικασία του χωρισμού αναπεριφέρειες. Αυτή η στρατηγική, η στρατηγική που παραθέτουμε στην ε, ιστοσελίδα μας, η οποία αναθεωρείται πολλές φορές, ορίζει τρεις ζώνες. Η μία είναι η πρόσφατα προσβληθεί στις περιφέρειες, όπως το Βέλγιο, από τον ιό. Και εκεί έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες που πρέπει να εφαρμόσουμε σαφής απαγόρευση μετατόπισης, μετα... Ε, για να κλειδώσουμε εκεί την αρρώστια. Επίσης έχουμε χώρες όπως η Στονία και η Λετωνία που ε, ήδη έχουμε κρούσματα και ε, ελάχιστος αγριόχειρους έχουμε ακόμη ζωντανούς γιατί έχουν προσβληθεί και θα πεθάνουν αλλά δεν μπορούμε να μειώσουμε τον πληθυσμό αγριοχείρων τόσο ώστε να εξαλείψουμε την όσο. Και επίσης έχουμε μια στρατηγική για τις ε, υγιείς περιοχές. Και εκεί που δεν έχουμε ακόμη κρούσματα θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό των αγριοχείρων και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη συνεργασία με τους κυνηγού. Και θα πρέπει οι κυνηγοί να αντιληφθούν τον ρόλο που παίζουν στο δάσος και στη διαχείριση ε, των αγριοχείρων. Είχαμε πάντως καλή συνεργασία μέχρι στιγμής με τους κυνηγού, θα πρέπει να αντιληφθούν και αυτοί γιατί θα πρέπει να κυνηγούμε συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί το ένστικτο του κυνηγού είναι να σκοτώνει τα αρσενικά και να μην σκοτώνει τα θηλυκά ζώα, ε, γιατί τα θηλυκά θα εξασφαλίσουν την διόνυση του πληθυσμού και άρα θα τους εξασφαλίζουν ε, θηρευτική περίοδο και του χρόνου, αλλά τώρα ε, έχουμε προσπαθήσει να διαπαιδαγωγήσουμε τους κυνηγούς για να μην κυνηγούμε τέτοιο τρόπο. Και θα πρέπει... Και μάλιστα έχουμε ξεκινήσει διάφορες εκστρατείες ε, ε, ενημέρωσης προς τις ε, συλλόγους κυνηγών για να τους πείσουμε ότι έχει στρατηγική σημασία η επιλογή της κυνηγητικής μεθόδου. Και αυτό το είδαμε και στο Βέλγιο. Εκεί ο εμπειρογνώμονο μας εξήγησε σε ένα μεγάλο ακροτήριο κυνηγών της περιοχής τι πρέπει να κάνουν και τι να αποφεύγουν. Και αυτό βοήθησε πολύ ε, να αποφύγουμε την περαιτέρω εξάπλωση της ζωνόσου. Και στο Βέλγιο προσπαθούμε να απομονώσουμε την αιστεία της ε, ζωνόσου για να μπορέσουμε να την ξεριζώσουμε την ε, επιζώτια και πολλοί αγριόχοι έχουν ε, είναι αντικείμενο κυνηγιού στα κρατημέλη και έγιναν ε, έλεγχοι για να δούμε αν είναι ε, άρρωστοι ή όχι. Πάντως, επαναλαμβάνω, το 99,5% του πληθυσμού αγριοχείρων θα ε, εξολοθρευτούν από την όσα. Από τη στιγμή που, μία, που η επιζωτία μπαίνει σε μία περιοχή, ε, είναι τελειωμένο το θέμα για τους αγριόχειρους. Δεν υπάρχει ε, πιθανότητα σωτηρίας. Σας ευχαριστώ. Ξεχάσετε με τις απαντήσεις ε, την πτήση που έχετε. Κύριε Χαϊταμα, μισό λεπτό και εσείς παρακαλώ. Μία ερώτηση μόνο. Άκουσα από τις ειδήσει ότι δεν έχουμε μόνο 12 κρούσματα στο Βέλγιο, αλλά 53. Είναι πολύ μεγαλύτερη έκταση από ό,τι είχατε no, φανταστεί. Είπα στην εισαγωγή ότι έχουμε πάνω από 50 αγριόχειρους που έχουν εντοπιστεί σε αυτή τη μικρή περιοχή με την επιζώτια. Και όλοι οι αγριόχειροι στην περιοχή θα ε, θα πεθάνουν. Δηλαδή την επόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι 100 και την επό, με την επόμενη 150. Το θέμα δεν είναι πώ είναι, είναι να μην φύγουν από αυτή την περιοχή οι αγριόχειροι. Γιατί ούτω ή άλλω όσοι αγριόχειροι βρίσκονται στην περιοχή θα πεθάνουν. Αλλά θέλουμε να, να απομακρύνουμε τα πτώματα του, τα σφάγια από, τη, από την περιοχή για να μην παραμένουν και να μολύνουν άλλα κοπάδια, γέλες αγριοχείρων που βρίσκονται σε γειτονικέ περιοχές. Πάντως, η συγκεκριμένη περιοχή που έχει ξεσπάσει ενώ όσους ε, ε, οι αγριόχειροι είναι καταδικασμένοι. Και δεν, από τη στιγμή που έχει φτάσει μία επιζωτία στην περιοχή, το αν το κρούσμα είναι ένα ή εκατό δεν έχει διαφορά. Επιδημιολογικά είναι ένα περιοριστή, είναι αναγκαίο να περιοριστεί σε συγκεκριμένη περιοχή η επιζωτία και να μην επεκταθεί σε γειτονικέ περιοχέ Και αυτό το χαρακτήρα έχουν τα μέτρα που έχουμε λάβει. Ο κύριο Καλινόφσκι. Ευχαριστώ. Συγγνώμη κύριε Διευθυντά. Είχα αποφασίσει να μην α, υποβάλω ερώτηση, αλλά είμαι υποχρεωμένος. Από τη μια λέτε ότι είναι αδύνατο να περιορίσουμε τον αριθμό των αγριοχείρων και από την άλλη λέτε ότι δεν θα μείνει ζωντανό ούτε ένα αγριόχειρο από τη στιγμή που έχει φτάσει η επιζώτια στην περιοχή. Τελικά τι θα γίνει. Ναι, Πρόεδρε στις ε, κάτω χώρες, στη χώρα μου, υπάρχει η επιλογή μηδέν. Ακριβώς για να μην ε, μολυνθούν οι κτηνοτροφικές μονάδες. Ε, δεν ξέρω τώρα αν αυτό ισχύει και για το Βέλγιο ή είναι κάτι παρόμοιο. σε, περιοχές που δεν έχουμε αγριόχειρους, όπως ας πούμε στη Δανία, στις κατοχώρες στο Βέλγιο, η ζωονόσος δεν θα επιμείνει. Μπορεί να επηρεαστεί, ας πούμε, μέσω ανθρωπινού ε, παράγοντα μια κτηνοτροφική μονάδα που μπορεί να επηρεαστεί, να μολυνθεί και θα χρησιμοποιηθούν τα, μέτρα που πρέπει για να σταματήσει η, ε, ε, η ασθένεια αν δεν έχετε ε, αγριόχειρο, λέμε πάντα. Μπορεί να εξελιχθεί η ασθένεια στις περιοχές που δεν υπάρχουν αγριόχειροι. Οι αγριόχειροι είναι που διατηρούν τον ιό για περισσότερο χρονικό διάστημα και βέβαια και στο περιβάλλον. Ο κύριος Καλινόφσκι. Α, όχι, συγγνώμη. Ε, ναι, γι' αυτό ακριβώς ρώτησα για την περίφραξη. Γιατί δεν έχουμε πολλούς αγριόχειρους. Και θέλουμε να τους εξοντώσουμε στη Δανία. Ελάχιστη είναι, θέλουμε να τους ξεφορτωθούμε. Και θέλουμε ε, να κάνουμε περιφράξεις ε, ε για να μην εισέρχονται οι αγριόχειροι στη Δανία. Γιατί είμαστε μεγάλη παραγωγή χείριου κρέατος. Αλλά η Επιτροπή λέει όχι μην κατασκευάσετε φράκτες. Πώς θα κρατήσουμε όμως τις περιοχές μας καθαρές από την Αφρικανική παρόλη των χείρων αν δεν κάνουμε περίφραξη για να μην μετακινηθούν προς εμάς οι αγριόχειροι. Ο κύριος Μπούντα. Ε, σε ό,τι αφορά την ταφή σε σχέση με την αποτέφρωση, δεν είναι καλύτερο να τους ε, καίμε αντί να τους θάβουμε ε, τους αγριόχειρους, τους νεκρούς αγριόχειρους. Νομίζω ότι είναι, μια και ο ιός μπορεί να παραμείνει ενεργός τρεις με τέσσερις μέρες, καλύτερα να τους καίμε παρά να τους θάβουμε. Ναι, ναι, ξέχασα τις δύο αυτές ερωτήσεις. Ό,τι αφορά την περίφραξη. Δεν λέω ότι είναι άχρηστος ο φράχτης. Απλώς ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Τροφίμων, ο ΕΦΣΑ, λέει ότι οι φράκτες σε μεγάλες αποστάσεις δεν προσφέρουν τίποτα γιατί θα βρει τρόπο αγριόχειρος να επιδείξει το φράχτη. Το έχουμε δει και στο παρελθόν με άλλες νόσους. Οπότε η περίφραξη δεν βοηθάει στον περιορισμό της νόσου. Τώρα, η εξολόθρευση του συνόλου των αγριοχείρων δεν γίνεται. Μπορεί να γίνει σε περιορισμένη περιοχή. Το κάναμε στη Ζεχία αλλά από τη στιγμή που έχουμε ένα μεγάλο δάσος, δεν μπορούμε να σκοτώσουμε όλους τους αγριόχειρους. Όπως δεν μπορούμε να σκοτώσουμε όλα τα, τα πτηνά που είναι φορείς τη ε, της ε, των πουλερικών, των πτηνών. Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε μηδενική παρουσία αγριοχείρων. Αλλά μηδενική παρουσία είναι απαραίτητη για να αναχαιτήσουμε την επέκταση τη νόσου. Αλλά αυτό όμω δεν γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να ζήσουμε με την αρρώστια αυτή. Σε ό,τι αφορά την ταφή, τα, τους διάφορου τόπου διαχείρισης ε, ε, των ασφαγίων υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Υπάρχει τρόπος ε, για, καθα... για καθαρή εξάλληψη των σφαγείων για λόγους βιοσφάλειας. Η καύση είναι ένας τρόπος. Θα πρέπει να λάβουμε μέτρα ώστε να αποφεύγεται η παρουσία του ιού στο, στο σφάγιο μετά την ταφή. Πάντως είναι αλήθεια ότι σε μερικές περιοχές και αυτό συνέβη σε πολλά κρατημέλη όταν έχουμε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων το πρόβλημα είναι υπάρχει ε, μεγάλος αποτεφρωτήρας ώστε να μπορέσει να καταστρέψει τεράστιο αριθμό σφαγείων. για παράδειγμα. Όταν είχαμε τον Αυθόδη Πυρετό στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρειάστηκε να θανατωθούν 8 εκατομμύρια ε, πρόβατα, υπήρχε ε, πρόβλημα με την ανέβριση τόσο μεγάλων εγκαταστάσεων για να πραγματοποιήσουμε την καύση, την αποτέφρωση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ήταν πολύ α, η παρουσίαση. Καλύπτεται και το παρελθόν και το παρόν. Η κυρία Αγγιλέρα μας υπεθύμησε ότι 35 χρόνια προσπαθήσατε να εξολοθρεύσετε αυτή την επιζώτια και τα καταφέρατε στην Ισπανία αλλά βιάζεστε, μου είπατε ότι έχετε αεροπλάνο, οπότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα για να προλάβετε και στην πτήση σας και να περάσουμε στο επόμενο θέμα, τα προβλήματα με τον ανταγωνισμό στον τομέα της γεωργίας. Έχουμε μία κρόαση με την παρουσίαση μίας μελέτης για την ΚΑΠ μετά το 2020 και τους νέους κανόνες για τον ανταγωνισμό. Ε, πρόκειται για μία μελέτη που θα βοηθήσει τον συντάκτη μας, τον ε, συγκεκριτή μας τον κύριο Ανδρείο που απουσιάζει όμως, ε, στα πλαίσια του μελλοντικού, της μελλοντικής κοινής οργάνωσης αγοράς και του σχετικού κανονισμού. Και επίσης να δούμε Πώ είναι οι κανόνε ανταγωνισμού, θα διευκρινιστούν και θα εδραιωθούν στη νέα ΚΑΠ, προκειμένου να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύση των γεωργών και των ενώσεων τους και ενώσεων παραγωγών. Ε, στα πλαίσια του κανονισμού Omnibus, ε, ε, θα έχουμε μια επισκόπηση του κανονιστικού πλαίσιου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ανταγωνισμό στα πλαίσια της ΚΟΑ και Έχουμε καλέσει εμπειρογνώμονες για το θέμα αυτό, την κυρία Κατρίν Τελκόντ, ε, που είναι καθηγήτρια στη Σχολή ε, Πολιτικών Επιστημών και Νομική Σχολή της Νάντς από τη Γαλλία και τον κύριο Αντώνιο Ιαναρέλη από το Πανεπιστήμιο του Μπάρι στην Ιταλία. Θα μας παρουσιάσουν οι δύο εμπειρογνώμονές μας τη μελέτη που τους αναθέσαμε και αν είστε έτοιμοι παρακαλώ Μπορείτε να ξεκινήσετε. 20 λεπτά έχετε συνολικά για την παρουσίαση της μελέτης. Και σας ακούμε για 20 λεπτά. Euh, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ. Okay. Les principaux points τα βασικά σημεία της μελέτης μας είναι τα εξής. Στόχος αυτής της μελέτης και στόχος της παρουσίασης είναι να αναφέρουμε εν συντομία τους ε, κανόνες ανταγωνισμού στη γεωργία και να σας γνωρίσουμε το νομοθετικό πλαίσιο όχι μόνο με βάση το θετικό, ε, τους θετικούς κανονισμούς αλλά και με τη βάση ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας προτείνουμε ορισμένες συστάσεις. Θα ήταν σκόπιμο να θυμίσουμε ότι το νομικό πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στη Γεωργία βασίζεται από το 58 από τη συνθήκη της Ρώμης στον πρωταρχικό ρόλο που παίζει η ΚΑΠ επί των κανόνων ανταγωνισμού. Το άρθρο 42 προβλέπει ότι αυτοί οι κανόνες ανταγωνισμού εφαρμόζονται μόνο ε, στην ε, εφαρμόζονται στον ε, εμπορία στο βαθμό που ορίζονται από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της κοινή αγροτικής πολιτικής και το άρθρο 39. Με άλλα λόγια, η ιδιαιτερότητα της γεωργίας και ο κοινωνικός ρόλος της ΚΑΠ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κανόνα των κανόνων ανταγωνισμού. Ε, το ευρωπαϊκό δίκαιο επιτρέπει να θυσιάζεται ο ανταγωνισμός προκειμένου να επιτευτούν οι στόχοι της ΚΑΠΑ. Με άλλα λόγια, στον γεωργικό τομέα η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού θα πρέπει πάντοτε να γίνεται με βάση τους στόχους της πολιτικής της ΚΑΠΕΠΗ του ανταγωνισμού, δηλαδή είναι καλύτερα να εφαρμόζονται οι κανόνες του ανταγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την οικονομική αποτελεσματικότητα του άρθρου 100 των συνθηκών, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του άρθρου 39. Από αυτό προκύπτει, όπως είναι λογικό, ότι οι πρακτικές αποφάσεις και η αποστολή των οργανώσεων παραγωγών και των οργανώσεών τους που ορίζονται από την κοινή αγροτική πολιτική είναι κατά ανάγκη εκτός του πεδίου εφαρμογής του ε, δικαίου ανταγωνισμού. Θα ήταν σκόπιμο να αναφέρουμε ότι αυτό ε, τονίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα Βάλε και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφαση της, ε, του 2017. Αναφέρεται σαφορητά ότι οι αποστολές ε, που αφορούν τις οργανώσεις των παραγωγών είναι, αποτελούν μία εξαίρεση του δικαίου ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά τις άλλες συμφωνίες και πρακτικές των παραγωγών και των οργανώσεων τους, υπόκειται στο άρθρο 101 της συνθήκης με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις που ορίζονται από το κανονισμό εφαρμογής της ΚΑΠΑ και με βάση τον κανονισμό από το 26-62 μέχρι τον κανονισμό του 13. Πράγματι, αυτοί οι κανονισμοί επιβεβαίωσαν την, τον ειδικό χαρακτήρα της προστασίας των ε, ε, γεωργικών παραγωγών γιατί όλες οι αποφάσεις που αφορούν αυτά τα προϊόντα δεν προβλέπονται από την εφαρμογή του άρθρου 101 επειδή πρόκειται για αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη στόχων του άρθρου 39 ενώ ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις οργανώσεις που κατά αποκλειστικότητα αποτελούνται από γεωργικούς παραγωγούς και οι οργανώσεις και οι συμφωνίες μεταξύ των παραγωγών που ε, ε, είναι ενταγμένοι σε οργανώσεις παραγωγών δεν καλύπτονται από την εφαρμογή του άρθρου 101 εκτός εάν υπάρχει αποκλεισμό ε, του ανταγωνισμού ή αν παρεμποδίζονται οι στόχοι της ΚΑΠΑ. Αυτή η διάταξη σύμφωνα με τη γεωργική πολιτική των τελευταίων δεκαετιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία μετά έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση, έθεσε όρια στη συμφωνία των παραγωγών. Οι συμφωνίες των παραγωγών σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να αφορούν τις γεωργικές τιμές ακριβώς γιατί οι γεωργικές τιμές ήταν διαρθρωτικό, συστατικό της γεωργικής πολιτικής. Λαμβάνοντα υπόψη αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε αυτό οδήγησε σε ορισμένους περιορισμούς σε ό,τι αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή αυτού του πλαισίου. Και από μία άποψη η υπεροχή των κανόνων της ΚΑΠ, η υπεροχή επί των κανόνων του αγωνισμού, κατά κάποιο τρόπο παραβιάστηκε και περιορίστηκε από την ερμηνεία που έγινε πρακτικά και από το δικαστήριο και από την Επιτροπή και ειδικά αυτό το πλαίσιο επιβεβαιώθηκε στον κανονισμό 1308 του 13 και η διαφορά μεταξύ όσων διέπονται από την ΚΑΠ και που ε, ε, ε, ε ερμηνεύονται στο άρθρο 206 στο οποίο γίνεται μία αναφορά στη συμπεριφορά των γεωργών με την επιφύλαξη των διατάξεων της ε, παρούσας ε, συνθήκης. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει μία αξιολόγηση με βάση τους κανονισμούς του ανταγωνισμού. Αντίθετα, αφο, ε, οι συμφωνίες μεταξύ παραγωγών καλύπτονται από τις συμφωνίες ανταγωνισμού. Ε, σε ό,τι αφορά την απαγόρευση ε, στον να επηρεάζονται οι τιμές εντάχθηκαν εδώ δύο εξαιρέσει. Η πρώτη εξαίρεση αφορούσε τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις για το γάλα που εισήχθησαν το 2011 και μετά αυτό επεκτάθηκε στα άρθρα 169, 170, 171 για τις διαπραγματεύσεις στον τομέα του ελαιόλαδου, ε, των δημητριακών και του βόηου κρέατος ενώ οι διατάξεις ε, για το γάλα ίσχυαν κατά αποκλειστικότητα με βάση ποσοτική ε, στοιχεία και σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο ευρωπαϊκό αντίθετα στα άρθρα 169, 70, 71 εισήχθη αυτή η εξαίρεση με βάση μία σειρά από προϋποθέσεις οι οποίες θύμισαν πολύ το κριτήριο της αποτελεσματικότητας της αγοράς ε, με παραπομπή στο 101 τρίτο εδάφιο. Δηλαδή υποχωρούσε η ΚΑΠ μπροστά στους κανόνες του ανταγωνισμού. Οπότε, ποιο είναι το κανονιστικό πλαίσιο για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού σήμερα μετά την έγκριση του κανονισμού Omnibus. Και ακριβώς μετά το πέρασμα α, μιας α, ε, ρυθμιζόμενης γεωργίας, σε μια γεωργία της αγοράς και με δεδομένη της αύξησης της ε, Δύναμη των αγοραστών εναντί των, παραγωγών, των παραγών, κρίναμε σκόπιμο να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική ισχύ των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, προκειμένου να ενισχύσουμε την ε, ισχύ των γεωργών στην, ε, στην αλυσίδα αξίας της γεωργίας και να καταπολεμήσουμε ταυτόχρονα τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Και μάλιστα η υπόθεση με τα κεχώρια έδειξε ότι ήταν αναγκαία μεγαλύτερη νομική ασφάλεια για τους οικονομικούς τελεστές σε ό,τι αφορά τον αποκλεισμό, την εξαίρεση, την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων και την θέση σε εμπορία των γεωργικών προϊόντων. Ο κανονισμός Omnibus περιέχει μια σημαντική τροπολογία ε, και της ε, κοινή οργάνωσης αγοράς, γιατί επεκτείνει την δυνατότητα συλλογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών ενοχικών διαπραγματεύσεων εκ μέρους των ενώσεων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών στο σύνολο των ε, προϊόντων και των παραγωγών. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτές οι συλλογικέ διαπραγματεύσεις μπορούν να αφορούν ταυτόχρονα και τις τιμές, κάτι που συνιστά αισθητή πρόοδο σε σχέση με τους όρους που ίσχυαν για τις τιμές στον κανονισμό 1308 του 2013. Έχουμε λοιπόν μία αναθεώρηση του νομικού πλαισίου εφαρμογής ε, του το δικαίου του ανταγωνισμού, των κανόνων του ανταγωνισμού και αυτή η τροπολογία είναι πολύ σημαντική γιατί όχι μόνο ενισχύει την υπεροχή της ΚΑΠ επί του ανταγωνισμού αλλά και ενισχύει τη θέση των οργανώσεων παραγωγών και ονώσεων οργάνων παραγωγών κατά τη ρυθμίση της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Το κείμενο αυτό αποτελεί σημαντική πρόοδο στην ε, ρύθμιση της ΚΑΠ. Σημαντική πρόοδος που αυξάνει την αποτελεσματικότητα της υπεροχής της ΚΑΠ και καθιστά πιο αποτελεσματικούς ε, τους στόχους της ε, ΚΑΠ, ενώ κατοχυρώνει την υπεροχή των στόχων αυτών έναντι του δικαίου ανταγωνισμού. Παρ' όλα αυτά, στον νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στη Γεωργία, θα πρέπει αυτό το νομικό πλαίσιο να εδραιωθεί και να διευκρινιστεί. Ε, χρειάζεται λοιπόν κατοχήρωση και διευκρίνηση αυτού του κανονιστικού πλαισίου για να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του νομικού κειμένου. Και από τη σκοπιά αυτή καταλήξαμε σε μια σειρά συστάσεων που γίνονται φυσικά με στόχο την εξασφάλιση ε, της υλοποίησης των στόχων της ΚΑΠ. Ο κανονισμός Omnibook ε, αντικατοπτρίζει τη σύγκρουση που προέκυψε μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής σχετικά με τη σχέση μεταξύ ΚΑΠ και ανταγωνισμού και αυτό είναι σημαντικό γιατί στην πρόταση μεταρρύθμιση της ΚΑΠ από πλευρά Επιτροπής το θέμα του ανταγωνισμού και το θέμα του ρόλου των οργανώσεων των παραγωγών δεν έτυχε προσοχή και δεν βρίσκεται στο κέντρο του θέματος. Στο κέντρο υπάρχει η προβληματική της συμμετρίας της, ε, στο εσωτερικό της όλης διαδικασίας. Αυτή η προβληματική όμως έχει μία επίπτωση σε επίπεδο νομικό και όχι σε επίπεδο ε, οικονομικό. Εκεί όπου μιλάμε για διαρθρωτική συμμετρία η απάντηση σε ό,τι αφορά την προστασία των συμβασικών σχέσεων αγγίζει ένα θέμα συγκυριακό ε, δευτερογενές σε ό,τι αφορά το κεντρικό χαρακτήρα των προβλημάτων που αφορούν κυρίως το θέμα που αυτή τη στιγμή μας απασχολεί. Ιδιαίτερα το θέμα αυτό και οι προτάσεις που γίνονται έχουν αναφορά στο άρθρο 152 της ΚΑΠΑ, όπως ε, μετά τις μεταρρυθμίσεις ε, του όμνιμπους γιατί κατά κάποιο τρόπο το θέμα είναι να πάψουν να υφίστανται ορισμένες αμφισβήμιες. Κατά την άποψή μας θα πρέπει να εξαλειφθεί η αναφορά στο άρθρο 101 που σήμερα περιέρχεται στο άρθρο 152 σχετικά με την διαπραγματεύσει των οργανώσεων παραγωγών, γιατί επειδή πρόκειται για ένα κανονισμό στο εσωτερικό τη ΚΑΠ η αναφορά σε αυτό το άρθρο είναι ανετιολόγητη παρά μόνο με βάση μια λογική που θα μπορούσε να αντιστρέψει ε, ε, ε, το θέμα της υπεροχής, της κάπα και της, ε, του ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες της οργάνωσης σχετικά με θέματα διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να εξαλειφθεί αυτή η αναφορά που γίνεται και που έχει σχέση με τις οργανώσεις για τις οποίες υπάρχει μεταφορά ιδιοκτησίας του προϊόντος, δηλαδή οργανώσεις οι οποίες συγκεντρώνουν την προσφορά και διαδραματίζουν ένα ρόλο και τις οργανώσεις που δεν ασχολούνται με αυτή τη συγκέντρωση και ε, δραστηριοποιούνται στις συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Το να βάζει κανείς μαζί αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι δημιουργεί αβεβαιότητες και υπάρχει κίνδυνος να πληγούν και οι συνεταιρισμοί οι οποίοι συγκεντρώνουν την προσφορά και ανέκαθεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν πολιτικές στο σχηματισμό των τιμών σε επίπεδο διαπραγματεύσεων δίχως να υπάρχει μια συγκεκριμένη άδεια σε ό,τι αφορά θέματα συμβιβασμού από την νομοθεσία. Τέλος, θα ήταν ε, σκόπιμο ε, λόγω της αναγνώρισης ε, του ρόλου που αποδίδεται από τον, την ομοθεσία σε οργανώσεις των παραγωγών να μην αποκλειστεί η δυνατότητα να υπάρχουν παρεμβάσεις από την Επιτροπή ή οργανώσεων παρι, αντιτράστα. Αλλά για να... οι ενδεχόμενες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να ισχύσουν για το μέλλον και να μην ισχύουν για το παρελθόν. Για όσα έχουν ήδη γίνει, μια τέτοιου είδους παρέμβαση ξεκίνησε στο Omnibus, αλλά χρειάζεται μια σαφέστερη ε, και συγκεκριμένη νομική λύση. Άλλες συστάσεις που κάναμε αφορούν το άρθρο 209 του κανονισμού για την ΚΟΑ. Το άρθρο αυτό αφορά τις εξαιρέσεις, δηλαδή τις συμπεριφορές που δεν εμπίπτουν στην κοινωνική πολιτική και δεν αποκλείονται άρα από το πεδίο εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού. Αυτό λοιπόν το άρθρο αφορά τις εξαιρέσεις. Το άρθρο 209 κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω, γιατί αφορά ταυτόχρονα με την παρούσα διατύπωση και τις ε, συμπεριφορές και τις πρακτικές και αποφάσεις των μη αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών, αλλά καλύπτει ταυτόχρονα τις συμπεριφορές ε, και αναγνωρισμένων ε, οργανώσεων παραγωγών που δεν εμπίπτουν όμως στις, στη νόμιμη αποστολή που προσδιορίζεται στο άρθρο 152. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να γίνει διάκριση ε, και προσδιορισμός του πεδίου ε, του άρθρου 209 ε, διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται στις μη αναγνωρισμένες οργανώσεις, αφενός και αφετέρου στις συμπεριφορές των αναγνωρισμένων ενώσεων οργανώσεων παραγών, που δεν εμπίπτουν όμως στον όρο των καθορισμένων αποστολών του άρθρου 152. Ε, και αν κάνω και πάλι παραπομπή στην υπόθεση για τα κεχώρια, το η υπόθεση αυτή ε, ε λύθη για τις συμπεριφορές που δεν έπτασαν στην νόμιμη αποστολή μπορούσαν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή του άρθρου 209. Και πάλι για το 209 άρθρο θεωρούμε σκόπιμο να καταργήσουμε την περίφημη ε, την, την απαγόρευση θεωρητρών του, του προσδιορισμού τιμών. Γιατί το άρθρο λέει ότι εξαιρέσεις δεν μπορούν να ωφελούν ε, αγο, ε, συμφωνίες με υποχρέωση προσφορά σε συγκεκριμένη τιμή. Και γιατί θέλουμε να καταργηθεί αυτή η απαγόρευση, γιατί είχε νόημα όσο υπήρχαν ρυθμισμένες τιμές. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που συνηγορεί υπέρ της κατάργησης, ε, της απαγόρευσης. Δεύτερον, ε, τέτοια απαγόρευση του price fixing δεν υπάρχει στο αμερικανικό δίκτυο και ε, η σχετική νομοθεσία που διέπει τα δικαιώματα των γεωργών στις ΗΠΑ από το 1922 ε, τους επιτρέπει να συνάπτουν συμφωνίες που εξαιρούνται από το δίκαιο ανταγωνισμού. Ακόμη και όταν εφαρμόζουν προσδιορισμένες τιμές. Τέλος θα έλεγα και πάλι υπέρ της κατάργησης της ε, απαγόρευσης ε, του προσδιορισμού τιμής, του price fixing, αν οι οικονομικοί τελεστές, οι παραγωγοί μπορούν να καθορίσουν κάποιες τιμές ε, και να συγκεντρώσουν την προσφορά, αυτό θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο άρθρο 172α που προβλέπει ε, ρήτρες ε, κατανομής της αξίας. Έτσι θα έχουμε καλύτερη κατακόρυφη διαπραγμάτευση σε όλη την αλυσίδα αξίας. Ε, και τελευταίο επιχείρημα που αφορά και πάλι την υπόθεση με τα Αυτό το νέο άρθρο 209 με τις δύο βασικές τροπολογίες θα έλυνε άπαξ και διαπαντός πρόβλημα που είχαμε στη διαμάχη με τα Κεχώρια που μας απασχόλησε για πολύ καιρό. Και κάναμε και κάποιες προτάσεις και στάσεις ό,τι αφορά την οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Και κυρίως την πρόταση για παράταση του πεδίου εφαρμογή, επέκταση του πεδίου εφαρμογή σε όλα τα γεωργικά προϊόντα και σε όλα τα τρόφιμα. Ε, και να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή και σε όλου του προμηθευτέ που είναι γεωργοί, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα γενικό ορισμό των αθέμητων εμπορικών πρακτικών και να, να περιλάβουμε μία μνήμη και της οικονομικής εξάρτησης των προμηθευτών. Αυτά, σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι τηρήσαμε το χρόνο που μας διαθέσατε. Σας ευχαριστώ. Όντως, μπράβο σας, τα καταφέρατε τέλεια. Ποιο το λόγο, ο κύριο Νταντάν πρώτα. Euh, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο και την ε, κυρία για την ε, ενδιαφέρουσα αυτή μελέτη. Θαυμάσιο ήταν το Σαββατοκύριακο που πέρασα ε, διαβάζοντάς το. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν γνωρίζει κανείς όλες τις λεπτομέρειες να δει με τις αναλύσεις. Θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση. Τελειώσαμε τις ε, διαπραγματεύσεις του Όμνιμπου στις 12 Οκτωβρίου, δηλαδή πριν ε, να γνωρίζουμε την, μελέτη, την ε, έκθεση του δικαστηρίου. Αν τα πράγματα είχαν ακολουθήσει μια άλλη σειρά θα μπορούσα να είχα γράψει κάτι άλλο. Παρόλα αυτά κρατάω αυτό που γράψατε ότι θα πρέπει να υπάρχει, ε, να καταβάλει κανείς σε μία Ηράκλειο προσπάθεια και από την άλλη πλευρά ε, να προσπαθήσει να ξεφύγει από αυτό. Θα ήθελα να κάνετε μερικά σχόλια σχετικά με τα όσα είπατε. Πιστεύω ότι επί της ουσίας της πρότασης σε ό,τι αφορά το άρθρο 52 γίνεται μία αναφορά στους ε, κανόνες ανταγωνισμού. Μιλάμε για μία ε, συγκεκριμένη επιλογή που έγινε από το συνομοθότη. Θα πρέπει κανείς ε, να αναλογιστεί τι ήταν η ΚΑΠ της δεκαετίας του 60. Θα έπρεπε τότε να εμποδίσει κανείς, ε, ε, κανείς οποιονδήποτε να, να παρέμβει με μια πολιτική τιμών. Όταν άλυξαν οι, όταν άλυξε ε, η, πολιτική αυτή πτυχή δεν άλλαξε και σήμερα η επιθυμία του Κοινοβουλίου είναι να προσαρμόσει την ε, πολιτική που αφορά τις παραγωγών σε αυτή την εξέλιξη μια αγοράς που είναι πλέον μια ελεύθερη αγορά και που τιμές καθορίζονται μετά από διαπραγμάτευση. Δηλαδή η διαγραφή στο άρθρο 100 έχει σχέση με μία νομική βάση και έχει σχέση μεταξύ των κυρώσεων, ε, ε, ε, υπάρχει διαφορά μεταξύ των ε, ε, κυρώσεων και των εξαιρέσεων. Σε επίπεδο πολιτικό, ε, η εξαίρεση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αν λάβουμε υπόψη τους παραγωγούς και όσου εμπλέκονται εδώ σε ό,τι αφορά τη μεταφορά του ιδιοκτησιακού καθεστώτο, θα μπορούσε να είναι ένα στοιχείο διευκρίνηση που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην επόμενη οργάνωση της αγορά. Γιατί εδώ το Omnibus διευκρινίζει εντελώς το θέμα αυτό τη μεταφορά ιδιοκτησία και της εξαιρέσεις που συνεπάγεται. Θα θέλω να σα επιβεβαιώσω ότι οι των αρχών ανταγωνισμού επιβεβαιώθηκε. Επιβεβαιώθηκε ότι αυτές οι αποφάσεις αφορούν το μέλλον. Πραγματικά υπάρχει σαφής βούληση του Κοινοβουλίου και θα πρέπει να το δούμε αυτό στα εκτιμώντας, γιατί στα εκτιμώντας ε, του κειμένου γίνεται ρητά αναφορά σε αυτό που είπατε για να θεωρηθεί ότι είναι ένα σημείο εκκίνησης και προστασία για το μέλλον. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 209, το άρθρο αυτό αυτό, όπως υπογραμμίσατε, έχει λειτουργικό χαρακτήρα, ο οποίος δεν έχει επιτευχθεί εντελώς και κατά συνέπεια χρησιμοποιείται περιορισμένα. Γι' αυτό το λόγο θα θελήσαμε να εφαρμόσουμε αυτό το προληπτικό μέτρο που θα μπορούσε να αφορά την υποβολή ενός προγράμματος και όχι την επιβολή μιας κύρωσης. Σε ό,τι αφορά την ιδέα της απέναδιαμόρφωσης του 209 θα πρέπει να γίνει μια εκτενής εξέταση γιατί δίχως άλλο τίθεται το θέμα του λειτουργικού χαρακτήρα αυτής της εξαίρεσης και τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνεται η εξαίρεση στο άρθρο 152 που είναι ρητή. Ακόμα και αν οι γαλλικές αρχές το 2018 έκαναν μία ερμηνεία σε ό,τι αφορά αυτό το κείμενο. Η, καταστο... η διαγραφή της ρήτρα των τιμών είναι ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω. Δεν, δεν ξέρω αν αυτό θα μπορούσε να απασχολήσει την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Αυτό το θέμα δεν έγινε δεκτό από τα μέλη τα άρθρα 159 και 142 δεν θα πρέπει να αμπληθούν και ενδεχομένως θα πρέπει να διερευνήσουμε την έννοια της ελάχιστης τιμής. Τέλος, σε ό,τι αφορά το άρθρο 209, αυτό είναι ένα σημείο που δεν έγινε δεκτό στην τριημερή συνάντηση του 2013, Υπήρχαν ε, οι γνωστοί συνδιαπραγματευτές και η Εστονική Προεδρία έδειξε μεγάλη κατανόηση. Σε ό,τι αφορά το 222, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μερικά από τα μέτρα 222 αφορούν δράσεις που είναι δράσεις σε διεπαγγελματικού ε, αμυγός ε, διεπαγγελματικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση σας. Ε, γίνεται την κατάλληλη στιγμή. Δίχω άλλο εμείς θα σκεφτούμε περαιτέρω αυτή την εξέλιξη του δικαίου ανταγωνισμού και όπως είπατε και εσείς έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στην γεωργική πολιτική. Έξι λεπτά ε, κάνετε, κύριε Νταντά, για την ανακεφαλαιότητα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί ο συνάδελφος Νταντέν ε, με πρόλαβε. Καταρχάς, ε, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εμπειρογνώμονες που καλέσαμε σήμερα. Όσοι, σαν και εμένα, έπαιξαν κάποιο ρόλο στον κανονισμό Omnibus, εδώ τώρα πολύ περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις ε, αθέμητες πρακτικές. Ε, τα όσα λέτε ακούγονται πολύ ευχάριστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα διάφορα επιχειρήματα που ελπίζω ότι θα μας βοηθήσουν κατά τη διάρκεια των δύσκολων διαπραγματεύσεων που όπως γνωρίζετε Ε, έχουν υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο, τα ψηφίσαμε με ευρύτατη πλειοψηφία και τώρα βέβαια είναι θέμα του Συμβουλίου με την βοήθεια της Επιτροπής που βρίσκεται εδώ και πιστεύω ότι αυτή η μελέτη θα μπορούσε να καταστήσει ακόμα πιο αποτελεσματική την εργασία των ε, κοινωτικών θεσμικών οργάνων προκειμένου να τελειώσουν αυτές τις τριμερείς συναντήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα ήθελα να προσθέσω αναφερόμενος περισσότερο στην Επιτροπή και όχι σε εσά. Με αυτά τα αποτελέσματα, με μία περαιτέρω επιστημονική μαρτυρία, όπως αυτή τη μελέτη, της μελέτης σας, σε ό,τι αφορά την επέκταση των προϊόντων και το θέμα της, του αθέμητου ανταγωνισμού και ιδιαίτερα της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε όλες τις επιχειρήσεις ε, σύμφωνα με την αρχή ότι το αθέμητο είναι αθέμητο, δεν είναι θέμα ε, οικονομικών διαστάσεων, δεν θα έπρεπε σε αυτό το σημείο η Επιτροπή να υποστηρίξει στεναρά αυτό που ψήφισε το Κοινοβούλιο και να μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο επί αυτών το σημείο και να ολοκληρωθούμε με τρόπο θετικό. Ευχαριστώ. Αυτό μου αρέσει. Ο κύριος Ντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ του ε, δύο εκπροσώπου ε, που ε, έκαναν την παρουσίαση. Δεν είμαι νομικός εγώ, ένα σημείο μόνο θέλω να σχολιάσω, γιατί τα υπόλοιπα τα, τα είπαν οι συνάδελφοι. Το θέμα των αγοραστικών κοινοτήτων. Νομίζω ότι δεν εκφράζεται, δεν εκφράζομαι απολύτω σαφώ. Μιλώ για τις αγοραστικέ κοινότητε στην Γερμανία, όπως α πούμε η 11. ο Παόλο Ντεκάστρο στο διαπραγματεύσει ε, στον τριμερή διάλογο. Νομίζω ότι θα το ξεκαθαρίσει αυτό. Αλλά επειδή έχουν δημιουργηθεί έτσι κάποιε ανησυχίε, ε, γι' αυτό το λέω. Δεν ε, υπήρχε πρόθεση να δημιουργήσουμε δυσκολίε για αυτέ τι κοινότητε, αλλά γνωρίζουμε επίση ότι στην Ευρώπη υπάρχουν και ενώσει όπου οι πολιτές ε, πρέπει να έχουν την ε, έδρα τους ε, στην, ανάλογα με την χώρα στην οποία θέλουν να πουλήσουν. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε ισότητα όπλων στον ανταγωνισμό και εδώ να πω το εξής. Άμεσα πρέπει να διαπραγματευτούμε και αυτό είναι σαφές. Εγώ είμαι μέλος του ΕΛΚ, της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του Κοινοβουλίου και όταν στην ομάδα μας συζητούσαμε το θέμα αυτό πριν από δύο χρόνια, ομόφωνα αποφασίστηκε ότι ναι, πρέπει να διαπραγματευτούμε. Έχουμε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης μέλη, στις ε, σκανδιναβικές χώρες, οι συνάδελφοι από τις χώρες ε, αυτές είναι πολύ φιλελεύθεροι σε ό,τι αφορά την οικονομία και ε, συμφώνησαν και αυτοί ότι ναι, χρειάζεται, υπάρχει ανάγκη διαπραγματεύσεων. Ελπίζω το αποτέλεσμα θα είναι καλό και οι γεωργοί αλλά και οι μεταποιητές θα μπορέσουν να ενισχυθούν σε αυτή τη μεγάλη αλυσίδα. Αυτό είναι ο στόχο άλλωστε και ελπίζω να τον πετύχουμε. Εγώ είμαι 14 χρόνια μέλο του Κοινοβουλίου και έχω ζήσει διάφορες παρεμβάσεις ε, στον τομέα αυτό το 2015 το 2005 είχαμε πει ότι θα, κατα... καταργηθεί το roaming και αυτό ήταν ένα σημάδι για την αγορά, ήταν σημαντικό γιατί οι μεγάλες εταιρείε δεν ήταν ε, ε, ε, διατεθειμένες να μειώσουν ή να διαθέσουν συμβόλαια σε καταναλωτέ για άλλες χώρες, οπότε φαίνεται κάθε φορά πότε είναι απαραίτητη παρέμβαση στην αγορά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ροπέ. Έχουμε και άλλους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τους καλεσμένους εμπειρογνώμονες για την παρουσίαση που μας έκαναν, τις μελέτες τους. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πολύ επίκαιρο άλλωστε. Έχω μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Ωραία λέξη ο ανταγωνισμός, αλλά έχω την αίσθηση ότι τον χρησιμοποιούμε για να προστατεύσουμε τους μεσάζοντες και τους ε, εμπόρους, τα σούπερ μάρκετ, τις αλυσίδες διανομής, ενώ αυτούς πρέπει να προστατεύσουμε είναι οι γεωργοί και οι καταναλωτές. Οι παραγωγοί που παρέχουν την πρώτη ύλη είναι ανυπεράσπιστοι και υφίστανται τους κανόνες μερικές φορές. Επιβάλλουμε κανόνες που τους φέρουν σε δυσμενή μεταχείριση σχέση με τους υπόλοιπους κρίκους αλυσίδα αξίας. Άλλοι καθορίζουν α, τις τιμές για τους παραγωγούς, όχι οι ίδιοι παραγωγοί. θα έπρεπε λοιπόν να προβλέψουμε κάποιο κατόφλι τουλάχιστον ότι, ώστε ένας γεωργός που κάνει επενδύσεις να μπορεί να κάνει προβλέψεις και να γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει, αλλά θα μπορέσει να επιβιώσει με τη δραστηριότητά του. Αν αφήσουμε λοιπόν ανήμπορο και ανυπεράσπιστο τον παραγωγό, τον γεωργό, θα χρειαστεί αργότερα να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα. Φυσικά, ε, Κάθε χώρα αντιμετωπίζει διαφορετική κατάσταση. Σε μερικέ χώρε το 20% των παραγωγών είναι οργανωμένοι, είναι μέλη συνεταιρισμών, ενώ σε άλλε χώρε 60% των γεωργών είναι μέλη συνεταιρισμών ή οργανώσεων παραγωγών. Και σε ό,τι αφορά τι επιδοτήσει έχουμε διαφορέ τη τάξη 30 με 40%. Όλα αυτά. Θα πρέπει να διορθωθούν θα πρέπει να, υπά... να... να αξιοποιούνται το ίδιο οι άμεσα ενισχύσεις από όλους και να, να ευνοούν τους πάντες. Τι νόημα έχουν οι άμεσε επενδύσει, μετά από ένα χρόνο χρεοκοπήσει ο Γιώργος. Οι τιμέ του γάλακτο είναι επίση άλλο πρόβλημα. Εκεί υπάρχουν τεράστιες διαφορές στις τιμές. Μερικές φορές οι τιμές είναι και τριπλάσια σε κάποιες χώρες από τις άλλες. Ποιο φταίει γι' αυτό, ποιο φταίει για αυτέ τι τεράστιε διαφορέ, οι κανόνε ανταγωνισμού ή τίποτα άλλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς έχουμε μια, ένα φεστιβάλ για γεωργικά προϊόντα στη χώρα μου και οι παραγωγοί μου είπαν ότι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα για να έρθουν σε επαφή με τους γεωργούς και με τις ε, συνεταιριστικές οργανώσεις για να εκπροσωπέσουν τα συμφέροντά τους. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη για να υπάρξει κινητοποίηση των γεωργών να μπουν σε τέτοιου είδους ενώσεις. Γιατί πολλές φορές αυτό είναι και η επιβίωσή τους στην αγορά. Στην ε, Ρουμανία έχουμε τέτοιες ε, συλλογικέ καλλιέργειες, είχαμε κομμουνιστικό καθεστώς και πολλές φορές πολλοί φοβούνται να μπουν σε ένα τέτοιο καθεστώς. Πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιο τρόπο να πιέσουμε τα κρατη για να μπορέσουν και αυτά να πιέσουν τους γεωργούς τους να ενταχθούν σε τέτοιες ενώσεις. Τώρα, για το θέμα των ε, τιμών που πουλούν οι ε, γεωργοί τα προϊόντα τους. Στην Ρουμανία είχαμε μια αύξηση της αγοράς των καυσίμων. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μηχανισμούς για να μπορέσουμε να προσαρμόζουμε τις τιμές στο τι γίνεται στην αγορά. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους εμπρογνώμονες. Δεν ξέρω αν είναι η Γενική Διεύθυνση ε, Γεωργίας ή η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού που είναι εδώ έξω εκπρόσωποι της Κομισιόν. Καλό θα ήταν να έχουμε και απαντήσει από τη Γενική Διεύθυνση ε, Ανταγωνισμού. Βλέπω ότι όλοι εμιδιούμε. Νομίζω ότι αυτή η Γενική Διεύθυνση διευθυνση ανταγωνισμου βλεπω οτι ολοι μιδιουμε νομιζω οτι αυτη η ε, βασική ε, Εσεί έχετε απόψει, εμεί συμφωνούμε με τι απόψει σα, αλλά δεν νομίζω ότι συμφωνεί και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για την πολιτική για τη γεωργία. Μπορείτε να μα δώσετε κάποια ιδέα για το πώ μπορούμε αυτή τη μάχη να την κερδίσουμε, γιατί προ το παρόν ο αγώνα είναι αμφίροπος. Ε, ακούσαμε τις, ε, τα όσα μας είπατε για τις αθέμεντες εμπορικές πρακτικές, αλλά εγώ θα ήθελα μια καθοδήγηση, γιατί αυτό το θέμα είναι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό που απορρέει δηλαδή από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, ότι η τιμή ε, υπερισχύει στο το επίπεδο του, καταναλωτή, χωρίς όμως να δίνεται καμία σημασία στα υπόλοιπα βήματα της ε, αλυσίδας ό,τι αφορά την ε, πολιτική για τη γεωργία. Σας ευχαριστώ. ε, κανονικά στην αρχή τη συζήτηση πρέπει να εγγράφονται οι ομιλητέ για να ξέρω πόσο χρόνο έχουμε και να το μοιράσω δίκαια. Αν στην πορεία ζητάτε το λόγο, αναγκάζομαι να σα περιορίσω. Αν από την αρχή ξέρα πόσοι ομιλητέ προβλέπονται στο κατάλογο, θα έκανα κατά αναλογία πιο δίκαιη κατανομή του χρόνου. Αλλά αν στην πορεία το δηλώνετε, τι να σα κάνω, κύριο Φλάναγκαν. Ε, Ευχαριστώ. Προχωράει η συζήτηση και όλο μας έρχονται νέες ερωτήσεις στο νου. Είναι πολύ ζωντανή η συζήτηση. Δεν είναι στατική, γι' αυτό έρχομαι ε, σχεδόν στο τέλος. Δεν ε, ήθελα να πω κάτι μέχρι να ακούσω την κυρία Μαγκίνες. Για πρώτη φορά συμφωνώ με την κυρία Μαγκίνες. Θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να ακούσω οι άνθρωποι της Κομισιόν τι έχουν να πούν για τα θέματα αυτά, γιατί όντως αυτό το σημείο είναι θεμελιώδους σημασία για την επιβίωση από, στην περιοχή που, από την οποία προέρχομαι εγώ και πολλοί συνάδελφοι. Όπως είπε και ο κύριος ε, ε, δεν είναι νομικός, εγώ, αλλά αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να φτάσουμε σε μια, σε μια κατάσταση όπου οι γεωργοί παίρνουν για την παραγωγή του δίκαιε τιμέ. ποιοι είναι οι κανόνες που μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ό,τι πρέπει να γίνει πρέπει να γίνει. Θέλω λοιπόν μια κατάσταση όπου μπορώ εγώ να πάω στο σούπερ μάρκετ και βλέποντας τις τιμές του προϊόντος, να μπορώ να καταλάβω πόσα πήρε ο γεωργός. Αν δεν, έχω, αν δεν ικανοποιηθώ, θα μπορούσα να πάω σε ένα άλλο μαγαζί και να ψωνίσω από εκεί και να πιέσουμε λίγο μέχρι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι ε, επιχειρήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά όλα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Σε ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον, ε, στον κύριο Μαγγέλε που είναι ο αναπληρωτής ε, γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη κρίμα που δεν έχουμε εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον αναπληρωτή διευθυντή της Γενικής Διεύθυνση Γεωργία, ο κύριος Μέγκελε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να πω καταρχάς ότι είμαστε χωρισμένοι σε γενικές διευθύνσεις αλλά η Επιτροπή μιλάει με μία και μόνο φωνή. Είναι διοικητικό αυτό και ε, μπορούμε να συντονιστούμε και το κάνουμε. Συνεπώς ε, θα προσπαθήσω να σας πω τις απόψεις της Επιτροπής σχετικά με τα θέματα που ετέθησαν. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι το θέμα που θέτουμε είναι όχι αν θα πρέπει να θυσιάσουμε τον ανταγωνισμό στο βωμό της γεωργίας, αλλά το αντίθετο. Το ερώτημα είναι πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων του γεωργικού τομέα, όπως εκφράζονται στις συνθήκες, και των ωφελών που θα μπορούσε να έχει ο ανταγωνισμός σε αυτό το συγκεκριμένο κλάδο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ότι υπάρχει μία προτεραιότητα, θα μπορούσα να πω, για την ε, γεωργία σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό. Το δικαστήριο όμως είπε σαφώς στην απόφαση του ότι η γεωργία δεν είναι μία περιοχή στην οποία δεν παίζει ρόλο ο ανταγωνισμός. Στην ουσία αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία κινούμεθα γιατί λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα όσα λέει το δικαστήριο. Και αυτό αντικατροπίζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν αυτά τα μέτρα τα τελευταία 20-25 χρόνια. Τώρα, το Omnibus αναφέρθηκε δύο-τρεις φορές, ε, όπως και ο κύριος Ντεκάστρο, είχα τη χαρά να πάρω μέρος στις τριμερείς ε, συνομιλίες που διήγησαν στο συμβασμό. Και θυμάμαι πολύ καλά ότι η συζήτηση αυτή ήταν ε, ιδιαίτερα πολύπλοκη και οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα που ικανοποίησε όλα τα μέρη, μόνο ότι η Επιτροπή χρειάστηκε να κάνει μία δήλωση. Είπαμε δηλαδή ότι θα επιθυμούσαμε να προηγηθεί μία αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα εξέταζε διάφορα θέματα κοινωνικά, γεωργικά κτλ. Το αποτέλεσμα ήταν ένα νέο άρθρο 152 που όπως είπατε δεν βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το 209 αλλά αυτό είναι η συνέπεια αυτού που συμβαίνει αν μια νομοθετική διαδικασία είναι ε, αυτόρμητη και θέτει ορισμένα θέματα που θα πρέπει λεπτομερώς εκ των προτέρων να, να ε, αναλυθούν. Είναι σημαντικό λοιπόν όταν ξεκινάμε αυτές τις συζητήσεις, οι συζητήσεις αυτές να γίνονται πάνω σε μια πολύ, με βάση μια πολύ λεπτομερή ανάλυση που αποκαλούμε ε, αξιολόγηση επιπτώσεων. Αυτό ήταν στην εφαρμογή το, την 1η Ιανουαρίου του 2018, τώρα είμαστε στον Οκτώβριο, δηλαδή ούτε καν 10 μήνες αργότερα. Δεν είχαμε κάποια εμπειρία πρακτική με το άρθρο, δεν υπάρχει νομολογία σχετικά με αυτό το άρθρο και πραγματικά συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Νταντέν ότι καταρχάς θα πρέπει να αποκτήσουμε κάποια εμπειρία, κάποιες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτού του άρθρου. Γιατί δίχως άλλο υπάρχουν μερικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από αυτό το άρθρο. Δεν είναι αναγκαίο σε ό,τι αφορά ορισμένα ερωτήματα για, για να, υπάρξει, να υπάρξουν άλλες κρίσεις, αλλά αυτό ακριβώς είπε ο κύριος Νταντέν. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ένα-δύο ε, θέματα. Έγινε μία σύσταση στη μελέτη να διαγραφεί αναφορά στο άρθρο 101. Νομίζω ότι αυτό είναι από τα θετικά αυτού του άρθρου, γιατί στην ουσία ελέγχει τις ε, επιπτώσεις των σχετικών διατάξεων. Τώρα γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία το άρθρο 101 δεν θα ισχύει. Ξέρουμε ότι στο παρελθόν, το ξέραμε στο παρελθόν και διαγράφοντας τώρα το μέτρο θα αναρωτούμε γιατί ο νομοθέτης δεν θέλει να ξεκαθαρίσει τις επιπτώσεις αυτές όταν υπάρχει το άρθρο 206 το οποίο λέει ότι ισχύουν οι κανόνες του ανταγωνισμού στο γεωργικό κλάδο. Μπορώ να συμφωνήσω και με κάτι άλλο που είπε ο κ. ότι δεν θα ήταν καλή ιδέα να επανέλθουμε και πάλι σε αυτή τη φάση. Άρθρο, το άρθρο 209 ε, αναφέρθηκε εδώ και πάλι. Πιστεύω ότι δεν είναι πλέον ε, κατάλληλη στιγμή για να επανέλθουμε εδώ. Αυτό θα πρέπει να γίνει με βάση μια ολοκληρωμένη ανάλυση των, ε, του 152 και 209. Η Επιτροπή, από ό,τι γνωρίζω, μέχρι στιγμής δεν εκλήθη να δώσει οποιαδήποτε ερμηνεία σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 209 και ενδεχομένω θα ήταν σκόπιμο να περιμένει κανείς ε, την Επιτροπή να ε, φέρει άποψη πριν να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί το άρθρο. Έγινε η πρόταση να διαγραφεί ε, η αναφορά η ρήτρα στον καθορισμό των τιμών. Αυτή δεν είναι πλέον κατάλληλη στιγμή για να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες ερμηνευτικές, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει μια ρήτρα καθορισμού των τιμών. Αυτό που απαγορεύει το μέτρο είναι να υπάρχει υποχρέωση επιβολής της ίδιας τιμής. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό ε, αν αυτό είναι ο καθορισμός των τιμών ή θα πρέπει να ερμηνευτεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να διευκρινίσουμε ε, πριν να ξεκινήσουμε δύσκολες νομικές διαπραγματεύσεις για αυτά τα μέτρα. Μερικά σχόλια για τα UTP, είπατε κυρία Ντεκάστρο, για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Εμείς αναφερθήκαμε σε αυτά τα επιχειρήματα πολλές ε, φορές. Ε, μπορώ να απαντήσω με τα επιχειρήματα που έχω χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν. Καταρχάς έχουμε πάρα πολλές ανησυχίες και το συζητήσαμε το θέμα αυτό στην Ειδική Επιτροπή και με τις νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου ότι τέτοια διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής θα ήταν πάντα από το άρθρο 43 της ε, ε, συνθήκης παράγραφος 3 ε, και αυτό είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ ολιστηρό έδαφος και δεν θα πρέπει να υπάρχει ο κίνδυνος να υιοθετήσουμε μία νομοθεσία που μετά από μερικούς μήνες θα θεωρηθεί, θα κριθεί άκυρη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεύτερον, η πρότασή μα διέπεται από την αρχή της επικούρικότητα και της αναλογικότητας, επικούρικότητα, γιατί πιστεύουμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση που υπάρχει νομοθεσία από 20 ε, χώρε μέλη δεν είναι καλή ιδέα να ε, νομοθετήσουμε ε, για σημαντικές πτυχές, αλλά να δώσουμε την δυνατότητα να προωθήσουν τα ε, όσα ήδη υπάρχουν. Αναλογικότητα σημαίνει ότι δεν θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις που δεν απαιτούν ρύθμιση. Ας πούμε, ε, μεγάλες εταιρείε λιανικού εμπορίου και πολυεθνικούς ε, διανομής ειδών διατροφής. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Εμείς προσπαθήσαμε το αμβλύνουμε αυτό κάνοντας αναφορά σε έψιλον. Ενδεχομένω υπάρχει και κάποια άλλη δυνατότητα να τραβήξει κανείς ε, μία διαχωριστική γραμμή. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που εξετάσαμε προσεκτικά. Ε, αφορά τις άδειες αγοράς, ε, τις συμμαχίες ε, ε αγοραστών. Ε, δεν πιστεύουμε ότι ο τρόπος αντιμετώπισης τους είναι η απαγόρευσή τους. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσον υπάρχει ανάγκη προκειμένου να προφυλαχτούν οι γεωργοί να ασχοληθούμε με συμμαχίες που γίνονται μεταξύ των μεγάλων παικτών της διατροφικής αλήσου. Αλλά αυτό θα τεθεί κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Και ο κύριος Ροπέη έθεσε το θέμα του γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στις τιμές των προϊόντων. Αυτό έχει σχέση με την κατάσταση της αγοράς. Δηλαδή αν η αγορά είναι πλεονασματική, αν είναι ελληματική, συνήθως ε, στις ελληματικές αγορές οι τιμές είναι υψηλότερες. Ε, αυτό έχει σχέση με την, ε, τον ανταγωνισμό στο κράτος μέλος και όπως είπατε και εσείς αυτά, τα, αυτά ποικίλουν σε ορισμένες χώρες μέλη η ύπαρξη ε, οργανώσεων παραγωγών και συνεταιρισμών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Υπάρχουν άλλες χώρες μέλη που ε, οι γεωργοί δεν κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Και αυτό βεβαίως επηρεάζει και τον ανταγωνισμό και έχει ε, ε στη μέσα. Ολοκληρώνοντας θα να πω ότι ήταν ιδιαίτερα καρποφόρες οι συζητήσεις που αφορούσαν τον κανονισμό Omnibus. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να επανέλθουμε σε όλα αυτά τα θέματα και να τα ξανανοίξουμε. Οι γεωργοί έχουν ένα, μια σχετική βεβαιότητα Τώρα το να τα ξανανοίξουμε και πάλι αυτά θα μας οδηγήσει στο να κινηθούμε προς την αντικατεύθυνση και θα καταστρέψουμε την ε, ε, σαφήνεια που επιτύχαμε τον 17. Ε, Αλλά βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας για περισσέρω συζήτηση αυτών των θεμάτων και να πρόκειται στο Κοινοβούλιο να αποφασίσει τι θα πρέπει να συμπεριλάβει στις ε, τροπολογίες για την ε, κοινή οργάνωση της αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση, παρόλο που το θέμα είναι εξαιρετικά δύσκολο και δύσκολο είναι να βρούμε ικανοποιητική λύση για όλες τις πλευρές. Είναι μάλλον ανέφικτο να προσβλέπουμε σε τέτοια λύση που θα ικανοποιεί τους πάντες. Ένα δεκάλεπτο μας έμεινε για τους εμπειρογνώμονες μας. Σας αρκεί, ελπίζω να σας αρκεί. Θα ήθελα να εκφράσω μερικές σκέψεις σε γενικού χαρακτήρα. Θα ήθελα να πω ότι με λυπεί το γεγονός ότι το άρθρο 39 που είναι ο πυλώνας της γεωργικής πολιτικής που για πολλές δεκαετίες συνδέθηκε με μια πολιτική τιμών, έκανε ρητή αναφορά στους γεωργικούς παραγωγούς για να μπορέσουν να έχουν ένα κατάλληλο εισόδημα και στους καταναλωτές για να έχουν τις κατάλληλες τιμές. Δηλαδή, στην ουσία το 57 λαμβάνονται υπόψη τα πιο αδύναμα μέρη, τα πιο αδύναμα σκέλη τους καταναλωτές και τους παραγωγούς. Η πολιτική των ποινών για, δεκαετί, για δεκαετίες βασιζόταν ε, στον συνυπολογισμό της μέγι, των μέγιστων τιμών στις περιοχές που υπήρχε έλλειψη και των ελάχιστων εκεί που υπήρχε πληθώρα. Υπάρχει, υπήρχε λοιπόν μηχανισμό ισορροπία. Ποιο είναι το πρόβλημα. Από τη στιγμή που έπεψε να υφίσταται η πολιτική των τιμών, η οποία περιέργω πώ ήταν μια πολιτική τιμών που αναγνώριζε, που ε, ε, αναγνώριζε ε, την αρχή του ανταγωνισμού γιατί ήταν πολιτική η τιμή. Σήμερα που η τιμή δεν είναι πολιτική θα πρέπει να, έχουν οι ενδιαφερόμενοι την εξουσία να διαπραγματευτούν. Η αναφορά που έκανα προηγουμένως το 1922 δεν είναι τυχαία, γιατί από το 1922 ο κανονισμός αυτός επιτρέπει στις οργανώσεις παραγωγών να ορίζουν την τιμή. Αυτό σημαίνει ότι στο, ανταγωνιστικό, στο δίκαιο ανταγωνισμού για τη γεωργία αναγνωρίζεται η ανάγκη για το δεδομένο αυτό. Ένα άλλο δεδομένο θα ήθελα να αναφέρω. Ενδεχομένω θα μπορούσε να φανεί περισσότερο τεχνικό, επιτρέψτε μου όμως να το υπογραμμίσω. Στην ε, απόφαση με βάση το προϋπάρχον κείμενο του κανονισμού Omnibus, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι μία οργάνωση παραγωγών θα μπορούσε να υιοθετήσει ακόμα και περιοριστικές αποφάσεις παραγωγής γιατί αυτό ήταν μέρος των καθηκόντων που είχαν αναγνωριστεί ως στόχοι ε, που νομιμοποιούσαν τις οργανώσεις. Μετά το Omnibus η ίδια αυτή η δραστηριότητα υπόκειται στην ίδια ρύθμιση των τιμών και θεωρείται ως εξαίρεση στο άρθρο 101. Όπως βλέπετε σε ό,τι αφορά το σημείο αυτό έγινε ένα βήμα προς τα πίσω, όχι ένα βήμα προς, γιατί αυτό που θα μπορούσαν οι οργανώσεις να κάνουν πριν και το αναγνώρισε και το ίδιο το δικαστήριο, τώρα μπορούν να το κάνουν στο εσωτερικό τους με αυτές τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από το 152 στη νέα του εκδοχή και όλα περνάνε ως εξαίρεστη στο 102. Υπάρχει δηλαδή μία ε, αντιστροφή. Στο παρελθόν υπήρχε η ΚΑΠ και το δικαστήριο έλεγε ότι δεν είναι ε, ε, εξαίρεση Τώρα ο κανόνας είναι ΚΑΠ, αλλά περιέργως πως στο εσωτερικό της ΚΑΠ λέμε ότι αυτός ο κανόνας ισχύει γιατί είναι ε, εξαίρεση από το 101 που σημαίνει ότι ο σεβασμός του ανταγωνισμού είναι ο βασικός κανόνας και η ΚΑΠ είναι ένας τρόπος για να παρεκκλίνει κανείς από τον κανονισμό. Το 48 όμως μας λέει ότι η ΚΑΠ υπερέχει και το σύστημα που δημιουργείται τεχνιέντος είναι ένα σύστημα που επιτρέπει, ε, παραδίδει τις ε, ε, οργανώσεις γιατί αυτό που μπορούσαν να κάνουν στο παρελθόν ως κάπο μπορούν να το κάνουν ως εκχώρηση της, του ανταγωνισμού. Εγώ ως νομικός δεν μπορώ παρά να το υπογραμμίσω αυτό. Βεβαίως οι πολιτικές επιλογές εναπόκεινται στους ε, νομοθέτες. Ε, Συμφωνώ απόλυτα με τον προλαλήσαντα. Θα ήθελα γενικώ να πω ότι έχουμε δει διαφορετικές ερμηνείες ε, και εμείς υιοθετούμε την νομική σκοπιά, τη σκοπιά του νομιμεθούς. Κατάλαβα αυτά που είπε ο κ. Μέγκελε, αλλά για το άρθρο 152 ε, και το άρθρο 209 υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Η διευκρίνηση του άρθρου 209 δεν θα επηρεάσει καθόλου την ερμηνεία ή την αντίληψη του άρθρου 152. Επίσης, ε, αν ρωτήσατε ποιο είναι η θέση του ανταγωνισμού και τι κάνει ο ανταγωνισμός. Εμείς δεν μιλήσαμε γενικά για τον ανταγωνισμό, αλλά για το δίκαιο ανταγωνισμό. Και νομίζω ότι είναι προς τιμήν της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης που έχει δύο σημαντικές πολιτικές την πολιτική ε, ε, γεωργία, κοινή γεωργική πολιτική και την πολιτική ανταγωνισμού, όπως ε, κατοχυρώνεται στο δίκαιο ανταγωνισμού. Και είναι τεράστια η συγκέντρωση δύναμης και τεράστια η διαπραγματευτική ισχύ των αγοραστών. Υπάρχει όμως ε, πολιτική και δίκαιο ανταγωνισμού. Καταρχήν ένα δίκαιο ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά τι δομές της συγκέντρωσης ε, και ένας έλεγχος της δεσπόζουσας θέσης και θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή ε, συνάρθρωση μεταξύ των διαφόρων πολιτικών τη Ένωση. Και δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ της κοινή γεωρικής πολιτική και τη πολιτική ανταγωνισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι αθέμητε εμπορικέ πρακτικές, στην πρόταση που υποβάλαμε δεν ζητήσαμε επέκταση του πεδίου εφαρμογή στο σύνολο των δικαιούχων, αλλά στους προμηθευτές. Στο σχέδιο οδηγίας προμηθευτές είναι η γεωρική παραγωγή και το θετικό δίκαιο, το συστικό δίκαιο της Ένωσης προσπαθεί ε, να καταπολεμήσει σε θέμα τις εμπορικές πρακτικές και η κακοπιστία ε, στο αρχικό δίκαιο ε, τιμωρείται σε όλες τις ένωμες τάξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή οδηγία, ό,τι και αν όποιο και είναι το πεδίο εφαρμογή, δεν μπορεί να τροποποιήσει τι διαρθρωτικέ αδυναμίε που υπάρχουν λόγω τη μεγάλη συγκέντρωση ισχύω στι αλυσίδε διανομή και γενικώ στην αλυσίδα αξιών. Ε, στην περίπτωση της Γαλλίας έχουμε την Amazon που συνάπτει συμφωνίες με τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και αντιλαμβανόμαστε αμέσω ε, την εύλογη ανησυχία των γεωργικών παραγωγών. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση ε, έχοντας δώσει το λόγο σε όλους τους ομιλητές. Ακούσαμε και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους εμπειρογνώμονες μας που δευτερολόγησαν. Οπότε μπορούμε να κηρύξουμε το πέρας της απογευματινής μας συνεδρίασης. Σίγουρα θα ξαναχρειαστεί να επανέλθουμε στο θέμα, αλλά εδώ είχαμε συζήτηση για τις νομικές διατάξεις, αυτό επικεντρωθήκαμε. Ευχαριστώ και μην ξεχνάτε αύριο ότι στις 9 θα ξεκινήσουμε με ψηφοφορίες και μην ξεχάσετε τις ηλεκτρονικές κάρτες σας για την ψηφοφορία. Καλό σας βράδυ.